Bonjour. Καλημέρα σας. Σας παρακαλώ καθίστε και κάνετε ησυχία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ευχαριστώ τα μέλη που είναι παρόντα. Σας ζητώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας και αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις και σχόλια θεωρούμε ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Το σχέδιο πρακτικών της, τετάρτης, της συνεδρίασης της 4ης και 5ης Δεκεμβρίου του 19 και της 20ης και 21ης Ιανουαρίου του 2020 είναι διαθέσιμα διαδικτυακά. Προτείνω να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά εκτός και αν ε, ε, διατυπωθούν ενστάσεις. Μέχρι αν δεν υπάρχουν στάσει, θεωρούμε λοιπόν ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα επισήμως και με μεγάλη χαρά να χαιρετήσω την άφηξη στις τάξεις της Επιτροπής μας τριών νέων συναδέλφων μετά το Brexit, η κυρία Ντέμπαρεκ, μέλος της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Σοφός, από το ID, ο κύριος Αλφονσί από την πολιτική ομάδα των Πρασίνων. Και έχουμε την κυρία Ζέμα, μη εγγεγραμμένη. Χαιρετίζω επίσης την παρουσία των αναπληρωματικών μελών, Κωσί Δεπουρνιού, κυρία Ντεπαρνιέ Γκρόνενμπεργκ, για ο, κύριος, ο πρώτος κύριος από το Ρινιού, η δεύτερη από τους Πρασίνους και ο κύριος Γκουσμάν. Ελπίζω ότι θα κάνουν πολύ καλή δουλειά στις τάξεις, στου κόλπου τη Επιτροπής μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερω που θα συνεργαστούμε με ε, ε, τα νέα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη. Γνωρίζω ότι, ότι σήμερα και αύριο γίνεται σύνοδος κορυφής έτσι ώστε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να επιδιώξουν να πετύχουν συμφωνία πάνω στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου έχει θέσει επιτάπητος μία πρόταση την οποία έχετε όλοι λάβει, εάν δεν απατώμε, και είδατε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αναφέρει και συμμερίζομαι πλήρως και ενστερνίζομαι πλήρως την άποψή του ότι η πρόταση αυτή του κύριου Μισελ είναι πάρα πολύ μακριά από τις επιδιώξεις μας και πολύ απέχει από τις ανάγκες της Ευρώπης για να χρηματοδοτήσει τόσο τις ιστορικές πολιτικές που εφαρμόζει όσο και τις νέες προτεραιότητες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Νταβίτ Σασόλη, έχει υπενθυμίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο από τον Νοέμβριο του 2018 να διαπραγματευτεί αλλά δεν είναι καθόλου έτοιμο να στηρίξει μια οποιαδήποτε συμφωνία με ένα οποιοδήποτε τίμημα. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, πιστεύω ότι θα συμφωνείτε όλοι ε, στο ότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε ικανοποίηση για ένα τόσο σφιχτό προϋπολογισμό, ο οποίος θυσιάζει την πολιτική συνοχής και παρουσιάζει πολύ σημαντικά κενά και ιστερήσεις. Μελετήσαμε σε βάθος και με τη δέουσα επιμέλεια την πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου και οφείλω να πω ότι η πρόταση του κυρίου Μισελ δεν είναι ούτε ισορροπημένη, ούτε ισότιμη, ούτε δίκαιη και ότι θέτει σε κίνδυνο την ε, σωστή εφαρμογή των στόχων συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού για την αξιοποίηση των διαφόρων ταμείων και κονδυλίων. Θα συνεχίσουμε να δρούμε σε αυτές τις ώρες που απομένουν μέχρι να συγκληθεί η η Σύνοδος Κορυφής ε, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ποιήση και αναλόγως με την έκβαση του Συμβουλίου αύριο θα σας αναφέρω τις αποφάσεις που θα κληθούν να πάρουν οι συντονιστές ε, με την ιδιότητα του μέλους και του συντονιστή στη δική μας Επιτροπή. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών λάβει ομοφόνος την απόφαση να αναστείλουμε τον τριμερή πολιτικό διάλογο μέχρι την σύνοδο του Φεβρουαρίου και ότι εν τω μεταξύ έχω επισήμως απευθύνει ε, επίσημη επιστολή στην Επίτροπο κυρία Ελίζα Φερέιρα ζητώντας από την κυρία Επίτροπο να μας προτείνει μεταβατικό κανονισμό για το έτος 2021, για αυτή την οικονομική χρήση. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Θα παρακολουθήσουμε με τη δέουσα επιμέλεια, με μεγάλη προσοχή, τα διακύβευμα, αυτό το οποίο θα διαμειχθεί εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Μια τρίτη παρατήρηση και ανακοίνωση έχει να κάνει με την αποστολή μας στη Σλοβακία. Ευχαριστώ τις πολιτικές μου ομάδες οι οποίες ε, μας έχουν ε, δώσει ονόματα εκπροσώπων και καλό τις υπόλοιπες που δεν μας έχουν στείλει ονόματα να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Το πρόγραμμα αφιερώνει σημαντικό μέρος ε, στο θέμα της δίκαιης μετάβασης των ανθρακοπαραγωγικών περιοχών και γι' αυτό το λόγο θα πάμε στη Σλοβακία, στην Πριβίτσα, στην περιοχή του Ορμένιτπρα και εκεί θα συναντηθούμε με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Είναι πολύ σημαντικό πέρα από τις συνήθεις επισκέψεις και αποστολές που, κάνει, που οργανώνει η Επιτροπή μας στις κατατόπους περιφέρειες και περιοχές, το πρόγραμμα των επισκέψεων να συνάδει με την ομοπαρασκευαστική επικαιρότητα, με την ομοθετική επικαιρότητα και γι' αυτό λοιπόν η αποστολή σε αυτή την ανθρακοπαραγωγική περιοχή θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη από τη στιγμή που εξετάζουμε το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Άρα πολύ σωστά τώρα ολοκληρώσαμε την ομαλή μετάβαση και μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που, το 4, που έχει να κάνει με την πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση του ε, Ταμείου για τη Δίκαιη μετάβαση. Η δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση επί της ουσίας. Το ΕΛΚ μου ανακοίνωσε το όνομα του εισηγητή. Πρόκειται για τον συνάδελφό μας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον οποίο χαιρετίζω και συγχαίρω και ο οποίος θα έχει μπροστά του να αναλάβει αυτό το βαρύ και σοβαρό καθήκον, να συνεργαστεί με το σύνολο των πολιτικών ομάδων για να καταλήξει στη βέλτιστη δυνατή πρόταση, ώστε το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο και όσο πιο ε, ε, πολύ αποτελεσματικό, με τις μεγαλύτερες δυνατές επιδόσεις. Γνωρίζω ότι το σύνολο των πολιτικών ομάδων, όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν κινητοποιηθεί ιδιαιτέρως για τον κανονισμό αυτό και έχουμε μπροστά μας μήνες κατά τους οποίους θα χρειαστεί να κάνουμε μια πολύ σκληρή δουλειά και ξεκινάει αυτή η πολύ σκληρή δουλειά από σήμερα το απόγευμα και γι' αυτό ε, θέλησα να προσκαλέσω με τη συνάντηση που είχαμε με την ε, Επίτροπο κυρία Λίζα Φερέιρα να προσκαλέσω, ε, να αξιοποιήσω αυτή την ορμή και αυτό το momentum για να ε, προσκαλέσω εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας κάνουν τεχνικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα έχουμε εργαστήριο για το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση που έχει οργανωθεί αυτό το εργαστήριο από το θεματικό τμήμα Π με δεδομένη την τεράστια σημασία που έχει αυτό το θέμα. Παρακαλώ να μην αποχωρήσετε από την αίθουσα, να μην φύγετε, διότι τα στοιχεία τα οποία θα μάθουμε από τις τεχνικές παρουσιάσεις σήμερα το απόγευμα θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και πολιτική θέση και άποψη. Θα αφιερώσουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα ε, τις εργασίες μας στο Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα για την Επιτροπή μας και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση είναι ένα νέο ταμείο, ένα καινούριο ταμείο το οποίο έχει τη φιλοδοξία να στηρίξει εδάφη, να στηρίξει περιοχές οι οποίες πλήττονται και θα πληγούν περισσότερο από αυτή τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Χαιρετίζω την Άννα Βάγνερ, η οποία είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη της αντίστοιχης μονάδας της Διεύθυνσης Στρατηγικής Διαχείρισης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εδώ για να μας παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Σας δίνω ευθύ αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Um, and thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ, ε, κύριε Ευρωβουλευτές, για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να σας κάνω την παρουσίαση και να παρακολουθήσω τη συζήτηση ε, που θα γίνει για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν. Είναι μια σημαντική ευκαιρία αυτή για μας και να παρουσιάσουμε το θέμα και να ακούσουμε ε, ερωτήσεις, απορίες που υπάρχουν για την πρόταση αυτή και η φιλοδοξία μας εδώ είναι να σας δώσουμε ε, μία ε, σε βάθος εικόνα ε, μετά από τις συζητήσεις που ήδη κάνατε με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Και σε σχέση με αυτό, ήδη ήθελα να σας πω πού εντάσσεται αυτό το δίκαιο, ε, το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση που εντάσσεται στο μηχανισμό δίκαιη μετάβασης που είναι η διάσταση η επενδυτική της πράσινη Συμφωνίας που παρουσίασε τον περασμένο Δεκέμβριο η Κομισιόν και που έχει την φιλοδοξία να κινητοποιήσει περίπου 100 ε, δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων, ε, ευρώ, με συγχωρείτε, επενδύσεων για τι περιοχέ που πλήττονται περισσότερο από την μετάβαση. Ο μηχανισμός δίκαιης μετάβαση που είναι ε, ένας ευρύτερος μηχανισμός από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι το ίδιο το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι το Ταμείο το οποίο θα ενταχθεί στην πολιτική συνοχής μαζί με τα άλλα ταμεία συνοχής και αναμένεται να δημιουργήσει επενδύσεις γύρω στα 30 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ παρέχοντας κυρίως επιχορηγήσεις. Ο δεύτερος πυλώνας του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, μετά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, είναι ένα ειδικό ε, πρόγραμμα ε, χρηματοδότησης που αποτελεί μέρος του προγράμματος Invest EU, που είναι ένα προϊόν που αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, ε, κυρίως προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και με τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων και της αγοράς επίσης. Τώρα, όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, ε, πρόκειται για μια δανειακή ε, διευκόλυση του δημοσίου τομέα στα πλαίσια του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, έχει, ε, ε, περιλαμβάνει μια διευκόλυνση δανειοδοτική που θα αναμένεται να δημιουργήσει γύρω στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο τρίτος πυλώνας έχει σαν φιλοδοξία να μοχλεύσει δημόσια χρηματοδότηση και απευθύνεται κυρίως σε φορείς του δημοσίου. Τώρα, α, αυτοί οι τρεις πυλώνες, όπως είπα, βρίσκονται κάτω από τον μηχανισμό ε, δίκαιης μετάβασης. Ένα βασικό εργαλείο για τη χρησιμοποίησή τους είναι τα σχέδια, ε, τα, εδαφικά ε, ε, σχέδια δίκαιης μετάβασης που θα προταθούν από τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή καταρτιστούν τα σχέδια αυτά από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς υπό την ευθύνη των κρατών μελών θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης και στους τρεις πυλώνες του μηχανισμού ε, δίκαιης ε, μετάβασης και ε, η ιδέα μας είναι ότι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας θα έχουν ευρύτερη θεματική και γεωγραφική κάλυψη με βάση τα εδάφη τα οποία θα έχουν προσδιοριστεί και εντοπιστεί μέσα στα σχέδια ε, ε, μετάβασης, τα οποία θα έχει εγκρίνει η Κομισιόν. Τώρα, ας περάσουμε στο τι φιλοδοξεί να κάνει αυτό το Ταμείο. Το πεδίο εφαρμογής και το αντικείμενό του. Το Ταμείο αυτό έχει σαν σκοπό να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα εδάφια εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης Προ μια ε, κλιματικά ουδέτερη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050. Το Ταμείο λοιπόν αυτό αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και όχι κατευθείαν ε, το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ε, το οποίο αντιμετωπίζεται μέσω ενεργειακών ε, προγραμμάτων και σχεδίων, όπως είναι, παραδείγματο χάρη, το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Αυτή η ιδέα όμως είναι ξεχωριστή, είναι κάτι το διαφορετικό. Και θέλω να το τονίσω αυτό το σημείο. Ο σκοπός μας είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που ε, η κλιματική μετάβαση θα έχει στα διάφορα εδάφη, στις διάφορες περιοχές των κρατών μελών και αναφέρεται αυτό στον ειδικό στόχο και στη διατύπωσή του. Ο ειδικό αυτός στόχος ε, αναφέρεται στον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της μετάβασης και παράλληλα με τον μηχανισμό δίκαιης ε, μετάβασης που είναι το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υπάρχουν και τα άλλα ε, μέσα της πολιτικής συνοχής, διότι το Ταμείο αυτό εντάσσεται μέσα στην πολιτική συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από τους κανόνες του κανονισμού κοινών διατάξεων που καλύπτει όλα, όλες τις πολιτικές συνοχές. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός κοινών διατάξεων θα καλύπτει τώρα και θα αποτελεί τους κανόνες και για το Ταμείο ε, Δίκαιης Μετάβασης. Τώρα, ποιοι είναι οι πόροι για το ταμείο αυτό. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, βασικά υπάρχει ένα ποσό 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ φρέσκου χρήματος, όπως λέμε, που προτείνει η Κομισιόν, ε, που ε, προστίθεται στο MFF του 2018, της, πρότασης του 2018. Ε, στο κεφάλαιο 3 προτείνεται να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση για την ενίσχυση των ε, δράσεων για τους ε, ε, φυσικούς πόρους και το περιβάλλον του MFF και αυτοί οι πόροι θα συμπληρωθούν μέσω υποχρεωτικών μεταφορών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι μεταφορές αυτές θα είναι τουλάχιστον μια μισή φορά ε, το ποσό που προτείνεται ε, για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και όχι πάνω από τριπλάσιο αυτού του κονδυλίου. Αυτό για να ε, τεθεί ένα πλαίσιο για, τις συνολικές, για τους συνολικούς πόρους που θα διατεθούν για το στόχο αυτό, επίσης και για να προστατεύσουμε τους πόρους της κοινωνικής συνοχής που χρησιμοποιούνται για την ε, για τους παραδοσιακούς στόχους της πολιτικής συνοχής για να αντιμετωπιστούν οι παραδοσιακές προκλήσεις, αν θέλετε να πούμε έτσι, της πολιτικής συνοχής και γι' αυτό ε, οι μεταφορές αυτές θα πρέπει να κρατηθούν εντός του 20% του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Κοινωνικού Ταμείου, ε, ώστε να υπάρχουν αρκετά κονδύλια και για τους σκοπούς των δύο αυτών ταμείων με έναν ισορροπημένο τρόπο. Τα ποσά τα οποία θα μεταφερθούν θα αιτιολογούνται στα εδαφικά σχέδια μετάβασης που όπως είπα έχουν κεντρικό ρόλο ε, στα πλαίσια της ε, υλοποίησης αυτού του ταμείου και το είδος των δράσεων που προβλέπονται ή που θα περιγράφονται σε αυτά τα σχέδια θα πρέπει να παρέχουν και ένα στοιχείο αιτιολόγησης για το λόγο για τον οποίο θα προτείνονται αυτές οι μεταφορές. Παραδείγματο χάρη, ε, Ο, αν υπάρχει μια πρόταση για να βοηθηθούν οι εργάτες που αναζητούν ε, θέσεις εργασίας ε, θα προέρχονται οι πόροι από το, ταμείο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η ιδέα επίσης των μεταφορών αυτών είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και ένα ενιαίο κορβανάς θα λέγαμε πηγή χρηματοδότησης για όλα αυτά τα μέτρα. Δεν θα υπάρχουν ε, πολλαπλά σύνολα κανόνων που να περιπλέκουν τα πράγματα. Θα υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Όσον αφορά τη δυνατότητα ε, μεταγενέστερης αύξησης των πόρων, υπάρχει αυτή η δυνατότητα που προβλέπεται σε κάποιο άρθρο Αργότερα, στα πλαίσια του MFF, οι πόροι μπορούν να αυξηθούν βάσει ε, αποφάσεων των δημοσιονομικών αρχών. Θα ισχύουν τα ποσοστά στη χρηματοδότηση όπως ισχύουν για την πολιτική συνοχής και πάλι ε, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν και για τις άλλες ε, πολιτικές συνοχής και τα άλλα ταμεία συνοχής, δηλαδή το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και το ε, Ταμείο περιφερικής Ανάπτυξης. Τώρα, ε, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες και δύο στόχοι που είναι η κινητήρια δύναμη της στήριξης αυτής. Από τη μία πλευρά προβλέπουμε να βοηθήσουμε τις περιοχές στις ε, ε, προσπάθειας τους μετασχηματισμού ώστε να διαφοροποιηθούν οι οικονομίες τους, να είναι λιγότερο ε, ευάλωτες και ε, να εξαρτώνται από τη μετάβαση αυτή. Και επίσης από την άλλη πλευρά ε, ένα μεγάλο μέρος των δράσεων αυτών θα εστιάζεται στην κοινωνική διάσταση της μετάβασης ε, με σκοπό να δοθεί υποστήριξη στους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να ε, αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και για να βοηθήσουμε με τον τρόπο αυτό τους αναζητούντες εργασία να ενταχθούν καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν ότι στο πεδίο εφαρμογής έχουμε στοιχεία και από το Κοινοτικό Ταμείο Πλάς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, υπάρχουν ε, δράσεις και των δύο ειδών που ε, πρόκειται να υποστηρίξουμε. Ε, επανέρχομαι στον μηχανισμό ε, δίκαιης μετάβασης. Το δεύτερο και τρίτο πυλώνα, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχει, έχουμε μια ευρύτερη τομεακή και γεωγραφική κάλυψη ε, με σκοπό να μπορέσουμε να καλύψουμε επεμβάσεις απαραίτητες και σχέδια τα οποία απαιτούνται για μια ε, επιτυχημένη ε, κλιματική δίκαιη μετάβαση. Το Ταμείο όμως δίκαιης μετάβασης με το, τα περιορισμένα κονδύλια που θα διαθέτει προτείνουμε να εστιαστεί μόνο σε κάποιους τομείς και να έχει ένα πιο περιορισμένο πεδίο ε, στήριξης. Όσον αφορά την ε, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η αηφορία και αυτό είναι το είδος επεμβάσεων ή έργων που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να ε, συμμορφώνεται πλήρως με την αρχή του ορυπένων πληρώνει» και όσον αφορά τα μέτρα εφορίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να τονιστεί η περιβαλλοντική διάσταση των περιοχών αυτών που κατά παράδοση υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχή με βάση κάποιους περιορισμούς. Όσον αφορά τους όρους επιλεξιμότητας ε, και πάλι τα σχέδια, τα εδαφικά σχέδια ε, δικές μετάβαση. είναι κεντρική σημασία για την επιλεξιμότητα των σχεδίων. Ε, θα πρέπει ε, να ε, υπάρχει σχέση με τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να υπάρχει ε, η κατάλληλη αιτιολόγηση στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης και οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στην ε, υλοποίηση των σχεδίων. Αν ε, μιλάμε τώρα για υποστήριξη σε συγκεκριμένα άτομα, αυτοί που θα υποστηρίζονται από το Ταμείο θα πρέπει αποδεδειγμένα είναι, να είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται από τις προκλήσεις που δημιουργεί η μετάβαση. Τώρα, πώς ε, δημιουργείται ε, το, το σύστημα επιλεξιμότητας στα πλαίσια αυτού του Ταμείου. Εδώ θα ήθελα ε, να τονίσω ότι συνάδει πλήρως σε γενικές γραμμές με τις επενδύσεις που είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πλάς. Αλλά εδώ υπάρχουν ιδιαίτερα δύο τομεί που θα μπορούσαν να πάρουν ε, πολύ περισμένες ε, επιπλέον επενδύσεις, δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και κάποιες δραστηριότητες υποστήριξης που έχουν σαν σκοπό τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά με πολύ αυστηρές προποθέσει που σχετίζονται με, τις, με την απώλεια θέσεων εργασίας ή με τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν στις, ε, στους τομείς αυτούς. Και μπορούν να αιτιολογηθούν αυτές οι επενδύσεις μόνο ε, με βάση την, ε, το λόγο ότι αντισταθμίζονται χαμένες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται θέσεις εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στα σχέδια και συνολικά θα πρέπει να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ε, ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Ε, σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού, και την αιρεσιμότητα. Η διαφάνεια αυτή συνοψίζει ένα βασικό ερώτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώς η πρόταση αυτή θα ενταχθεί στην ε, εξελίξη διαδικασία που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, ε, ε ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όταν το ε, συνολικό νομικό νομικό πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή όπως ελπίζουμε ε, στις αρχές του 2021, η διαδικασία προγραμματισμού θα έχει προχωρήσει ήδη αρκετά, ούτω ώστε τα, ε, οι προτάσεις να μπορούν να υποβληθούν ήδη στην αρχή ε, θέσεως σε ισχύ του νομικού πλαισίου και ήδη οι, πολύ γρήγορα οι δικαιούχοι να αρχίζουν να υλοποιούν. Όσον αφορά τη διαδικασία προγραμματισμού, η Κομισιόν έχει ανακοινώσει κάποια αναλυτικά στοιχεία ε, υπό τη μορφή των εκθέσεων αναχώρα και των ε, παραρτημάτων που ε, ε, ισχύουν για το Ταμείο ε, Δίκαιης Μετάβασης. Έχει κάποια στοιχεία η Κομισιόν τα οποία θα μοιραστεί με τα κράτη-μέλη στα τέλη αυτού του μήνα και ε, αναφέρονται εκεί αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ποια εδάφη απειλούνται περισσότερο και ποιε είναι αντίστοιχα οι προκλήσει. Αυτό είναι ένα ε, σημείο αφετηρίας ήδη για να, γίνουν κάποιες, ε, να ξεκινήσουν κάποιες ανεπίσημες συζητήσεις από τώρα για το μελλοντικό αυτό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που θα πρέπει να ενταχθούν και στο επίσημο πλαίσιο όταν θα προκύψει. Και όλα αυτά θα πρέπει να ε, ε, τροφοδοτήσουν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης ε, μετάβασης, τα οποία σχέδια όταν μιλάμε για το εθνικό επίπεδο πλέον και τις δεσμεύσεις που θα αναλυφθούν σε επίπεδο κρατικό ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και θα πρέπει να περνάνε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανάλυσης και λεπτομέρειας, ε, ούτως ώστε να είναι βέβαιο ότι καλύπτονται οι περισσότερο πληττόμενες περιοχές και επίσης ούτως ώστε να υπάρχει μια περιγραφή ανά ε, εδαφική περιοχή σχετικά με τα προβλεπόμενα ε, μέτρα, ε, τις συγκεκριμένες δράσεις που πρόκειται να ληφθούν, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ούτω ώστε τα σχέδια αυτά μέσω ενός επικοδομητικού διαλόγου να συμφωνηθούν μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών και τα σχέδια αυτά με τη βοήθεια του Ταμείου Δίκαιης ε, Μετάβασης να υιοθετηθούν τελικά. Και από αυτού θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι εφόσον το Ταμείο αυτό και ο προγραμματισμός του εντάσσονται πλήρως στο ε, πλαίσιο πολιτικής συνοχής, η συμμετοχή των εταίρων, των εταιρικών σχέσεων και ε, τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά σεβαστά ε, μέσω, σύμφωνα και με αυτά που βλέπει ο κανονισμός κοινών διατάξεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και την περιγραφή των ενδιαφερόμενων φορέων που θα εμπλακούν στα σχέδια ε, δίκαιης μετάβασης. Αυτό ε, είναι, είναι μια υποχρεωτική πληροφορία που θα πρέπει να περιλαμβάνεται για να ξεκινήσει ο σχετικός διάλογος. Όσον αφορά τη μέθοδο κατανομής, θα ήθελα να σας δείξω ποια είναι τα βασικά κριτήρια τα οποία ε, λάβαμε υπόψη μας όταν ε, προτείναμε την κατανομή και θα δείτε ε, εδώ ότι αναφέρονται τέσσερα, πέντε συγγνώμη, στοιχεία η μισή από τους δείκτες αυτούς αναφέρονται στην οικονομική πτυχή και στην, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των ε, εδαφών, των περιοχών για τις οποίες πρόκειται και το άλλο η μισή των δικτών αυτών, η άλλη μισή αναφέρονται και αντικατοπτρίζουν τις ε, προκλήσεις απασχόλησης που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτό το Ταμείο. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ε, βιομηχανικών εγκαταστάσεων ε, σε περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα και όσον αφορά την απασχόληση, έχουμε την απασχόληση στη βιομηχανία, την απασχόληση στην εξόριξη άνθρακα και λιγνίτη που λαμβάνονται υπόψη και επιπλέον έχουμε την παραγωγή τύρφης και την παραγωγή ε, πετρελαιού σχιστόλιθου με σκοπό να προσαρμοστούν ε, συνολικά όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ούτω ώστε να υπάρχει ένα στοιχείο αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης στην κατανομή αυτή και προς τις δύο κατευθύνσεις υπάρχει ε, ένα συνολικό ανώτατο όριο στις, ε, στα ποσά αυτά, ώστε ποτέ να μην ε, υπάρχει υπέρβαση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ένα κράτο και από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα όγκου χρηματοδότηση που λαμβάνει σαν ελάχιστο 6 ευρώ κατά κεφαλή καθ' όλη την περίοδο. Κάποιες ε, διορθώσεις επίσης εφαρμόζονται στη μέθοδο αυτή και αυτό με σκοπό να λαμβάνεται υπόψη το καθάριστο εγχώριο εισόδημα ε, κατά κεφαλή στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να ε, εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση των πόρων στα λιγότερο ενεπτυγμένα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή τη μεθοδολογία, το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στην οθόνη σας τι θα προκύψει δηλαδή, όπου εδώ βλέπετε όχι μόνο την κατανομή των κονδυλίων, αλλά βλέπετε και άλλες δύο στήλες που είναι τα ποσά που αναμένεται η Κομισιόν να κινητοποιηθούν μέσω του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος και του τρίτου πυλώνα που είναι η δημόσια ε, δανειοδότηση και η συμμετοχή επίσης της ΕΤΕΠ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την προσοχή σας ε, και φυσικά περιμένω να λάβετε ε, τη δέουσα υπόψη αυτή της, να δέλετε τη υπόψη σε αυτή τις προτάσεις όπως και με βέβαια θα πράξετε. Ευχαριστώ. Κυρία Βάγκνα, ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είχατε την βγαίνει να εδώ και θα σας παρακαλέσω να παραμείνετε μέχρι τέλους, να ακούσετε και τους εμπειρογνώμονες και μετά ξέρετε θα απακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και είμαι βέβαιος ότι θα σας τεθούν και εσάς προσωπικά πολλές ερωτήσεις. Θέλω να καλωσορίσω και τον αγαπητό τέο συνάδελφο Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι. Πραγματικά χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ Λάμπερτ που σε ξαναβλέπουμε και πολύ σύντομα θα είσαι εδώ, θα κάθεσαι εδώ, διότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να οργανώσουμε αυτή τη στιγμή είναι μια συνάντηση ε, στην οποία θα λάβεις εσύ υπόψη και σημαίνω και θα μας παρουσιάσεις τις κατευθύνσεις της πολύ σημαντικής οργάνωσης της ΕΣΠΟΥΝ που ε, στόχο έχει να προωθήσει τη συνοχή στην Ευρώπη. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Ε, θα ήθελα να δώσω καταρχάς ε, το λόγο στον δόκτωρα Βαγγέλη Τζίμα, τον πρώτο μας εμπειρογνώμονα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών έρχεται ο κύριος Τζίμας που θα μας μιλήσει για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των αυτοπαραγωγικών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο κύριε Τζίμα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Περιμένω λίγο το remote control. Αλλά καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και ε, τους βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας τα πορίσματα ενός πονήματος που έγινε στο κοινό κέντρο ερευνών ε, της Επιτροπής και αφορά τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν ε, στο πλαίσιο της μετάβασης για την κλιματική ουδετερότητα, ενθρακοπαραγωγικές ε, περιοχές, αλλά κυρίως να σας παρουσιάσουμε και τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες οι οποίες θα δημιουργηθούν, ιδίω για τη διατήρηση αλλά και την επέκταση, όπως θα σας δείξω, Τη απασχόληση και άλλων ευκαιριών σε περιφερειακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την οικονομική μεγέθυνση. Όσοι δεν γνωρίζετε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, είμαστε ένα κέντρο γνώσεων ε, και επιστημών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρέχουμε επιστημονικές ενδείξεις και αποδείξεις ε, και συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας ε, σε διάφορες γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2017 ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν περιοχε που εξαρτώνται από τον άνθρακα ε, στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια κλιματική ουδετερότητα και σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε για την ε, δημιουργία ενός πολύ ισχυρού εργαλείου για τη μετάβαση αυτών των περιοχών, ένα εργαλείο που θα τις υποστηρίξει, αλλά συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη παρέχοντάς τους ε, ε, τις απαραίτητες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τα απαραίτητα μοντέλα μέσω των οποίων ε, θα προχωρήσει αυτή η μετάβαση χωρίς να αντιμετωπίσουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τι κάνουμε λοιπόν. Καταρχάς προσπαθούμε να αντιληφθούμε τις προκλήσεις. Είναι σαφές ε, ότι η μετάβαση κλιματική ουδετερότητα ε, θα οδηγήσει σε απόσυρση των ε, δραστηριοτήτων αυτών και των υλικών αυτών. Έξι κράτη-μέλη ακόμη και σήμερα βασίζονται κατά πάνω από 20% για τις ανθρωπικές ανάγκες σε αυτά τα προϊόντα. Έχουμε, εξ γνωρίσουμε τουλάχιστον, 128 ανθρακοριχεία σε 12 κράτη-μέλη και 42 περιοχές ΝΑΤΣ2 που παράχουν ε, πάνω από 5 δις ε, τόνους ε, άνθρακα ή λιγνίτη που καλύπτει τα 3 τέταρτα της κατανάλωσης του 150 50 το 1 τρίτον ε, της συνολικής ε, ε, δυνατότητας καλύπτεται από τα εργοστάσια στις 21 χώρες. Βέβαια γνωρίζουμε ότι σιγά σιγά παρετούνται, εγκαταλείπουν αυτό το κλάδο τα κράτη-μέλη, από, συναρμολογούν, παροπλίζουν τις μονάδες αυτές από αυτές τις 8 που είπα το 2016 κατά ένα τρίτο κατά 100 δηλαδή ε, θα εγκαταληφθούν και θα μείνουν ε, πολύ μικρότερες. Βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά τα νούμερα. Την πληρέστερη εικόνα θα την έχουμε το καλοκαίρι οπότε και θα εκτιμηθούν τα εθνικά κλιματικά προγράμματα. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις περιφέρειες όταν θα παραμείνουν, όπως είπα, το 2030 περίπου 55 γιγαβατόρες. Βλέπετε πόσοι απασχολούνται στην Ένωση, 52.700 περίπου στα εργοστάσια. Αλλά έχουμε 185.000 ε, στις εξωτερικτικές δραστηριότητες που απασχολούνται. Βέβαια, το βάρος ε, είναι επιμερισμένο και όχι κατά ισομερή τρόπο. Είναι χώρες που θα ε, θυγούν περισσότερο και άλλες λιγότερο. Η Πολωνία, για παράδειγμα, 130.000 ανθρώπους απασχολεί άμεσα στον τομέα αυτό. Και θα πρέπει να προσθέσουμε και πάνω από 215.000 ανθρώπους οι οποίοι έμεσα ε, δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό, δηλαδή σε Συναφή παρεμφερή εργασία. Δηλαδή μιλάμε λίγο πολύ για μισό εκατομμύριο ανθρώπου που εργάζονται στον τομέα τη παραγωγή άνθρακα. Αν λάβουμε υπόψη τώρα και την απόσυρση και κατάληψη αυτών των μονάδων, θα υπάρξουν και σημαντικέ απώλειε θέσεων εργασία. Υπολογίζουμε 77.000 θέσει να έχουν χαθεί μέχρι το 2025 και 160.000 μέχρι το 2030. Είναι μια πρόκληση και θα πρέπει να δούμε όμως και τι ευκαιρίες μπορεί να διανοιχθούν και να προκύψουν από την όλη αυτή μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να βοηθηθούν οι περιφέρειες ε, να διέλθουν με δίκαιο τρόπο αυτή την περίοδο μετάβασης, να μην μείνει πίσω κανείς. Θέλουμε εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα για την ε, διατήρηση, ίσω και αύξηση των θέσεων εργασία και θέλουμε οι περιοχέ να έχουν τι δυνατότητε ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν έτσι περαιτέρω. Παρά την εγκατάλειψη του άνθρακα, έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά ενώ είναι γενική η πρόκληση, τοπικά και περιφερειακά θα βρεθούν οι λύσει. Κατά τον σχεδιασμό λύσεων και στρατηγικών μετάβαση για τι περιφέρειες αυτέ, λαμβάνουμε υπόψη και την κατάσταση εγκατάλειψης δηλαδή του άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων, αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο, τον αντίκτυπο στη κοινωνία, τον περιβαλλικό αντίκτυπο κτλ. Και θα πρέπει επίσης να δούμε πώς τα νέα εργαλεία, τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας, όπως νέες αλυσίδες ε, αξίας ή ψηφιακός μετασχηματισμός, πώς θα μας υποστηρίξουν ε, στο να βρούμε αυτές τις τοπικές λύσεις. Επίσης δεν υπάρχει μία ενιαία λύση η οποία να καλύπτει όλους τους τομείς και τι περιφέρειες, γιατί σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να βρεθούν οι πιο ενδεδειγμένε αναλλακτικέ προσεγγίσει, παράδειγμα χάρη με ξεχρονισμό άλλων κλάδων, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και να υπάρξουν και κάποια άλλα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προκληθούν με την ε, παράδοση που έχουν οι περιφέρειες και την έχουν αναπτύξει τόσα χρόνια που ε, εργάζονται ε, με τον άνθρακα. Άρα, πού θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στον άνθρωπο. Αυτό είναι σαφές. Και για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο τη απανθρακοποίηση, τη απαλλαγή από τον άνθρακα στην κατάσταση των ανθρώπων αυτών, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα σχέδια, ε, στρατηγικά σχέδια, καθώ και μια βαθμιδόν αναδιάρθρωση ε, στο βιομηχανικό κλάδο, ώστε να μπορούν ε, να προσαρμοστούν στη νέα οικονομία που θα προκύψει μετά την απαλλαγή από τον άνθρακα και την εφαρμογή τη Πράσινη Συμφωνία. Δεν θα πρέπει αυτέ οι περιοχέ να ξεκινήσουν από το μηδέν, έχουν κληρονομιά έχουν στοιχεία υπέρ τους, έχουν υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, αλλά ένα από τα βασικά τους ε, ατού είναι ο κόσμος ε, που δουλεύει εκεί, που έχει εξειδικευμένες δεξιότητες, ηλεκτρικές, μηχανολογικές, εργάζονται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, έχουν εμπειρία και πολύ μεγάλη και στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ άλλων, άρα είναι κατάλληλοι να απασχοληθούν σε άλλους τομείς όπως είναι οι εξορρυκτικές δραστηριότητες. Εγώ όμως θα εστιάσω ε, στη συνέχιση του επιχειρηματικού μοντέλου αυτών των περιοχών ε, στις, καθαρές ενέργειες, ε, στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, αιωλική, ηλιακή κυρίω. Ήδη υπάρχει μετάβαση σε αυτές τις περιοχές, ήδη υπάρχουν υποδομές παραδείγματος χάρη στον τομέα της ε, ηλιακής και ολικής ενέργειας για την εγκατάλειψη των ε, φραγκοριχείων και σε περιοχές που πριν υπήρχαν τέτοιες δραστηριότητες. Υπάρχει ανάπτυξη γης, υπάρχει πρόσβαση παραδείγματος χάρη σε δίκτυα υψηλή τάση ε, και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει και μεγαλύτερη αποδοχή από την κοινή γνώμη για αυτέ τι βιομηχανικέ εγκαταστάσει. Υπάρχουν και οι πόροι, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν νέε δεξιότητε για να μπορούν να βρουν ευκαιρίε και να απασχοληθούν σε εναλλακτικού κλάδου, όπω όπως, όπως είπα είναι οι τεχνολογίε καθαρή ενέργεια. Τι κάναμε την τελευταία χρονιά. Προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε το δυναμικό πράσινης ενέργειας σε 42 περιφέρειες που θα πληγούν. Αυτές οι περιοχές πρέπει να καταλάβουμε ότι θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό. Έχουμε κάνει κάποιους υπολογισμού για να δούμε ποιο είναι το τεχνικό δυναμικό ε, για τη βιοενέργεια, την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια σε περιοχές ε, που έχουν ανθρακοριχεία σήμερα. Δεν θα σας ζαλίσω με νούμερα γιατί μπορείτε να τη διαβάσετε στην έκθεση, έχετε αντίτυπα, μπορείτε να τα βρείτε στο βάθος της αίθουσας. Αυτό όμω που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά πρώτον υπάρχει δυναμικό ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας στι 42 αυτές περιοχέ περιοχές που θα καλύψει τουλάχιστον το μισό των ΑΠΕ που χρειάζονται για να καλυφθεί η φιλοδοξία της ε, απαλλαγή από τον άνθρωπο μέχρι το 2050. Και το βλέπετε και στο χάρτη. Αυτό το δυναμικό είναι διασπαρμένο στην Ευρώπη. Νότια Ευρώπη θα ωφεληθεί από την ε, ηλιακή ενέργεια σημαντικά, αλλά στο βορρά και στην Ανατολική Ευρώπη και από την αιωλική ενέργεια και τη βιοενέργεια. Άρα μπορείτε να δείτε ότι έχουμε δυναμικό, σημαντικό δυναμικό για μία διαφορετικές επιλογές και εναλλακτικέ. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι έχουμε σημαντικό δυναμικό και για τον εξυγχρονισμό ε, του υπάρχοντος εξοπλισμού και θα δοθούν νέες δυνατότητες και απασχόλησες, αλλά θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Ήδη στις περιφέρειες, τυπικά μέσω χαμηλής οδήματος, Τα κτίρια δεν καλύπτουν ε, τις απαιτήσει και με τον εξυγχρονισμό που γίνεται, με του τους που γίνεται θα χρειαστούν πάνω από 100 χρόνια για τον εξυγχρονισμό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον εξυγχρονισμό για να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση των κτηρίων, βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά έτσι δημιουργούμε και νέες θέσεις εργασίας, γιατί ανθρώπους που απασχολούνταν στον τομέα των ανθακορχείων θα τους απασχολούμε πλέον στον τομέα της οικοδομής, που είναι παρόμοιος κλάδος. Και θα πρέπει βέβαια να δούμε και πέραν των νεούσιμων πηγών ενέργειας και της τεχνολογίας που σας προανέφερα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχω εδώ είναι οι δυνατότητε απασχόλησης σε στα λεγόμενα giga factories για τους ορευτές που είναι πάρα πολύ απαραίτητοι για την κλιματική ουδετερότητα, για τη δική μετάβαση. Έχουμε και την ε, ηλεκτροκίνηση, θα μειώσουμε σίγουρα τα θερμοκηπιακά αέρια στον τομέα των μεταφορών που είναι ο πιο δύσκολο ω τομέα. Ε, ο κλάδο ε, έχει ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις ε, και τις παρακολουθούμε. Έχουμε τουλάχιστον 13 να έχουν προχωρήσει ήδη είτε στον τομέα του σχεδιασμού είτε και έχουν περάσει στο στάδιο της κατασκευής και πολλές από αυτές τι πρωτοβουλίες τι βλέπουμε σε θαρκοπαρογέ περιφέρειε. Για του σωρευτές ένα τέτοιο γιγαργοστάσιο μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας σε 3.000 ανθρώπους. Το δυναμικό αυτό πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε λοιπόν σε ευκαιρίες απασχόλησης. Αν πάρουμε υπόψη ε, τους πεφωνημένους στόχους ε, για τη μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030 που έχουμε στους στόχους και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε 315.000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ, αλλά και στις οικοδομές, ε, κατασκευή νεόδμητων ή ε, ανακαίνιση κτηρίων. 2.000 σήμερα είναι αυτοί που εργάζονται στις ίδιες περιοχές κατά αναπεριοχή. Άρα ε, θα έχουμε πολλαπλασιασμό των θέσεων εργασία, όχι ότι είναι ολαρόδινα βέβαια. Δεν θα ωφεληθούν όλοι το ίδιο από αυτή τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Και κοντεύω να κλείσω την παρέμβασή μου. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια τελευταία στοιχεία. Τι κάναμε μεταξύ άλλων Αφού είδαμε το δυναμικό σε κάθε περιφέρεια, προσπάθησαμε να υπολογίσουμε τι δυνατότητε ε, και τι ευκαιρίε δημιουργία νέων θέσεων εργασία με βάση αυτό το δυναμικό. Και έχουμε ομαδοποιήσει τι 42 αυτέ ε, περιφέρειε σε τρει διαφορετικέ οικογένειε. Έχουμε 28 ανθρωποπαραγωγέ περιφέρειε, πάνω από τι μισέ, οι οποίε έχουν πολύ ψηλό δυναμικό για την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Εδώ λοιπόν τι θα χρειαστεί. Να εξασφαλιστεί πω Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε αυτέ τι περιφέρειες. Έχουμε τώρα άλλε 7 περιφέρειες, μια δεύτερη ομάδα, όπου εδώ είναι παρόμοιο το δυναμικό, πολύ παρόμοιο με αυτό που ε, τώρα παρατηρείται ω προφίλ σε αυτέ τι περιοχέ, άρα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη υποστήριξη για να υπάρχει όσο δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση. Και υπάρχουν και δυστυχώ 7 περιφέρειες όπου το δυναμικό δημιουργία νέων θέσεων εργασία μέσα στον ΑΠΕ είναι πολύ χαμηλότερο από το υφιστάμενο επίπεδο απασχόληση στον τομέα αυτό. Ε, γι' αυτό χρειάζεται ξεκάθαρη προσπάθεια οι περιφέρειε αυτέ να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα εγκαταλείποντας τον άνθρακα και να ορίσουν ή να προσπαθήσουν να εξεύρουν απασχόληση και ανάπτυξη μέσω άλλων δραστηριοτήτων. Ολοκληρώνοντα, θα βρείτε στην έκθεσή μα και άλλε πολύ χρήσιμε πληροφορίε για τι περιοχέ επίπεδου ΝΑΤΣ 2. Θα δείτε πληροφορίε για κάθε τέτοια περιφέρεια το τεχνικό δυναμικό για τις διάφορες πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το δυναμικό ε, για τα κτίρια, την ανακαίνιση δηλαδή κτιρίων, το δυναμικό για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε υφιστάμενα ή εγκαταλειμμένα θρακορία και τέλο τι ευκαιρίε απασχόληση που έχουν δημιουργηθεί. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σα παρουσιάσω τα αποτελέσματα και ολοκληρώνοντα θα ήθελα να περάσω κάποια βασικά μηνύματα. Όπω είναι προφανέ οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας μπορούν να διευκολύνουν την ενεργειακή μετάβαση και να δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία. Με τέτοια έργα θα ε, στηριχθεί σίγουρα η περιφέρεια που ήδη έχει τις ακατάλληλες υποδομές, δεξιότητες, βιομηχανική κληρονομιά, στενή συνεργασία με εταιρείε, ρυθμιστές, επενδυτές, ε, χωροταξικούς σχεδιαστές, τοπικές κοινότητες είναι κάτι αναγκαίο για να εντοπιστούν οι πιο βιώσιμες χρήσεις. Βέβαια, θα πρέπει να βρεθούν και εναλλακτικέ δυνατότητε απασχόληση για ένα περιορισμένο αριθμό περιφερειών και βέβαια ο ενεργειακός τομέας είναι η μόνη λύση για τις περιφέρειες αυτές και θα πρέπει ε, να δούμε πού μπορούμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις και εκτός αυτού του τομέα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Τζίμα, για την παρουσίασή σας. Θα ακούσουμε τώρα τον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Ενρίκο Μπότα, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Θα μας ε, παρουσιάσατε την αναθεώρηση της στρατηγικής για τη διαχείριση της μετάβασης, προκειμένου να ε, πάμε σε μια οικονομική δραστηριότητα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, με χαμηλή ένταση άνθρακα. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και ένα τρίτο εμπειρογνώμονα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Μπότα, παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου, αλλά και για την παρουσία όλων εδώ. Είναι ένα εργαστήριο πολύ σημαντικό ε, γιατί το θέμα απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και ο σκοπός μας είναι να μάθουμε ο περισσότερο μπορούμε όλοι για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω μια μελέτη την οποία έχουμε εκπονήσει εντός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και προσπαθούμε να την φέρουμε σε πέρας με διαφορετικές ιδιότητες. Πρώτα, ε, προσπαθήσαμε να δούμε τι γνωρίζουμε για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, ποιους κλάδους θα πλήξει, ποιους εργαζομένους θα πλήξει. Μετά είδαμε προηγούμενες εμπειρίες από βιομηχανική μετάβαση και από αλλαγή της οικονομικής δραστηριότητας στο παρελθόν και είδαμε τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε και στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε ε, δίκαιες λύσεις για να φέρουμε σε πέρας, για να ε, διεξαχθεί ομαλά αυτή η μετάβαση. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το πρώτο μέρος της μελέτης. Έχει να κάνει με, το, με αυτά που γνωρίζουμε για τη μετάβαση προς χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και τη σχέση της με την απασχόληση. Φαίνεται να είναι σχετικά μικρό συνολικά ο αντίκτυπος. Αυτό, αυτή η μελέτη μιλάει για έναν υψηλό φορο άνθρακα, 50 δολάρια ανά τόνο, ενώ το σημείο αναφοράς είναι κυρίως 30 ε, δολάρια ανά τόνο, άρα βλέπετε ότι το, το νούμερο είναι ψηλό και με αυτή την παραδοχή ο συνολικός αντίκτυπος θα, θα, θα αντιστοιχίσει στο 0,2% αναπασχόληση. Ο συνολικό αντίπτυπος τι εννοώ με αυτό, όχι μόνο τις θέσει που θα χαθούν, αλλά και τις θέσει που θα δημιουργηθούν. Μιλούμε για ανακατανομή εργασιακή. Το 0,2% είναι πολύ χαμηλό νούμερο. Γιατί, διότι για παράδειγμα από το 1995 μέχρι το 2005, σε αυτή τη δεκαετία, κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΣΑ είχαμε ένα ποσοστό ανακατανομής θέσεων επασχόλησης ύψους 20%. Άρα καταλαβαίνετε γιατί μπροστά στο 20% το 0,3% φαντάζει ελάχιστο. Και γιατί φαντάζει ελάχιστο, φαντάζει διότι οι κλάδοι που επηρεάστηκαν δεν ήταν οι κλάδοι όπου οι εργοδότες ήταν οι μεγαλό... μεγαλύτεροι και οι εργαζόμενοι οι περισσότεροι. Κάποιοι κλάδοι θα πληγούν περισσότερο η εξορρυκτική βιομηχανία, τα διαφόρων είδων ορυχεία. Θα έχουμε 8% μείωση της απασχόλησης στον τομέα των ορυχείων και βλέπουμε και αλλαγή στον κλάδο των ενεργειακών της παραγωγικής ενέργειας, από την παραγωγή ενέργειας ε, με υψηλή ένταση άνθρακα σε παραγωγή ενέργειας με χαμηλή ένταση άνθρακα. Άρα το σημαντικό που πρέπει να κρατήσει κανείς από αυτή τη διαφάνεια είναι ότι η μετάβαση προς χαμηλή κατανάλωση άνθρακα πράγματι θα πλήξει διάφορους κλάδους, π.χ. τα ανθρακοριχεία και άλλους κλάδους υψηλής έντασης ενέργειας, αλλά δεν είναι μια διαδικασία καταστροφής θέσεων απασχόλησης, είναι μια διαδικασία μεταστροφής θέσεων απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι μετακινούνται από τον ένα κλάδο στον άλλο, καθώς χάνονται θέσεις απασχόλησης στον ένα κλάδο, δημιουργούνται σε κάποιον άλλον. Τι ξέρουμε λοιπόν για τους εργαζομένους σε αυτό ε, το κλάδο. Είναι μακριά η, οθόνη και έπρεπε να είχα φτιάξει μεγαλύτερες διαφάνειες. Ε, Κυρίως άνδρες τελεχώνουν την εξορρεκτική βιομηχανία. Θα είναι άνδρες ενήλικοι οι οποίοι θα πληγούν κατά κύριο λόγο από την μετάβαση αυτή. Η παραγωγή ενέργειας με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα είναι ένας οικονομικός κλάδος που δημιουργεί ευκαιρίες και για οικονομική ανάπτυξη αλλά και για απασχόληση. Οι γυναίκες παίζουν μεγαλύτερο ρόλο σε, στους κλάδους που παραδοσιακά κυριαρχούνται από άνδρες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες, γυναίκες είναι το 35% των εργαζομένων στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, ενώ γυναίκες είναι το 20-25% στις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Οι γυναίκες ήδη δουλεύουν σε αυτό το κλάδο ε, διοικητικά καθήκοντα εκτελούν και λιγότερο τεχνικά καθήκοντα ή καθήκοντα διοίκηση. Στο κλάδο δηλαδή όπου η παραγωγή ενέργειας έχει χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Αυτό συμβαίνει διότι οι γυναίκες ε, έχουν ε, ε, σε μικρότερο ποσοστό είναι πτυχιούχοι πολυτεχνείου και θετικών επιστημών που χρειάζεται τέτοιου είδους πτυχιούχους αυτή η βιομηχανία. Η επέκταση δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, προκλήσεις για τις γυναίκες, παρόλο που η μετάβαση και η εγκατάλειψη του άνθρακα θα πλήξει την ανδρική εργασία. Σε ορισμένες χώρες ε, οι εργαζόμενοι που πλήττονται είναι μεγαλύτερη ηλικία από άλλου. και αυτό ισχύει κυρίω για τι οικονομίε, για τα κράτη που είχαν οικονομίε με κεντρικό σχεδιασμό στο παρελθόν και που είχαν τέτοια ε, παράδοση. Είναι πιο δύσκολο για αυτούς να βρουν νέα θέση απασχόλησης για διάφορους λόγους είναι πιο απίθανο να συμμετάσχουν σε μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης. Ε, άλλωστε υπάρχει μεροληψία από τους εργαδότες και δεν τείνουν να προσλαμβάνουν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Αυτή η γραφική παράσταση είναι πολύ περίπλοκη να ε, γίνει αντιληπτή. Είναι δύσκολο να την καταλάβει κανεί και θα προσπαθήσω να σα την περιγράψω. Δεν είναι μονολόγο που, ε, το ότι είναι η οθόνη μακριά. Η μετάβαση θα επηρεάσει και εργαζομένου χαμηλών δεξιοτήτων και εργαζομένου υψηλών δεξιοτήτων. Δεν πρέπει κανεί να έχει υπόψη του ανθρώπου οι οποίοι είναι χειρονάκτε, είναι εργαζόμενοι με, λίγες, με λίγα προσόντα, ότι αυτοί θα πληγούν παραπάνω. Ακόμα και πολλοί προσοντούχοι εργαζόμενοι μπορεί να πληγούν. Θα χαθούν θέσει Απασχόληση σε ορισμένους κλάδους και θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης σε άλλους. η διαδικασία δημιουργίας θέσεων απασχόλησης θα είναι ε, ε, γρήγορη. Το σημαντικό είναι να έχουν τα σωστά προσόντα για να κάνουν τη μετάβαση εργαζόμενοι από το ένα κλάδο στον άλλο. Ποια προσόντα λοιπόν θα χρειαστούν. Αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο απασχολούνται πριν και από το πού θα βρουν δουλειά στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε τις ανάγκες. Για έναν ε, εργάτη ορυχείου πρέπει να μεταστραφεί προς τις κατασκευές ή προς τις επιχειρήσεις και το εμπόριο. Σύμφωνα με την προηγούμενη του εμπειρία, πρέπει να έχει κατάρτιση για να αναζητήσει αντίστοιχη θέση απασχόλησης. Και αυτό είναι σημαντικό στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, να εντοπίσουμε πιθανά, πιθανά μέρη στην αγορά εργασίας όπου μπορούμε να διοχετεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, μιλήσαμε λοιπόν για την απώλεια θέσεων ε, ε, απασχόλησης στην, στα ανθρακοριχεία και στην ανθρακοπαραγωγικό κλάδο, όμως Πρέπει να πούμε ότι ο ΣΑΧΙ έχει κάνει μελέτες σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και είδε ότι υπάρχουν διάφοροι κλάδοι μεταποίηση ε, σε, στη μεταλλουργία, ε, παραγωγή ε, οπτάνθρακα, Όλα αυτά ε, είναι δραστηριότητες που, είναι, ε, που βρίσκονται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και άρα σύσσωμη μια περιοχή μπορεί να πληγεί και είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή και πρέπει να την εξετάσουμε. Εάν πρέπει να μετακινηθούν οι εργαζόμενοι για να βρουν νέα θέση απασχόλησης, αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κοινότητα και στην οικογενειακή ζωή τους. Και επίσης η μεγαλύτερη σε ηλικία εξ αυτών που ήδη ε, είναι περισσότεροι σε αυτό το κλάδο, απλά θα αρνηθούν, μπορεί να αρνηθούν αυτή τη μετάβαση. Άρα η γεωγραφική απόκληση είναι κάτι το σημαντικό ε, και πρέπει να εξεταστεί. Τώρα, ε, αυτές είναι οι προκλήσεις. Ποιες είναι οι λύσεις. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω με λεπτομέρεια τις διαφάνειες αυτές. Να σας πω ότι Είδαμε τις εμπειρίες του παρελθόντος από την εξωρικτική βιομηχανία και είδαμε τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε. Έχετε τις πληροφορίες ε, στα δημοσιεύματά μας. Ε, οι περιπτωσιολογικές μελέτες όμως υπογραμμίζουν το εξής. Για να γίνει μια μετάβαση, το πρώτο που χρειάζεται είναι μακρόπνος, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Είναι μια μακρά διαδικασία. Η διαρθρωτική προσαρμογή σε αυτές τις περιοχές είναι κάτι που χρειάζεται μέχρι και 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όταν λοιπόν συζητούμε το όραμά μας, το ποιο μέλλον θέλουμε να σφυριλατήσουμε, είναι σημαντικό να εμπλέξουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, όλους τους φορείς. Στην Αλμπέρτα του Καναδά, όπου γίνεται ένα project αυτή τη στιγμή για τη δίκαιη μετάβαση, δημιουργήθηκε μια task force, μια ειδική ομάδα, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, εκπρόσωποι των εργαζομένων, να συμβάλλουν όλοι για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής, διατυπώνοντας προτάσεις. Άρα έχουμε στρατηγικές για την τοπική ανάπτυξη και πρέπει να βρούμε ε, θύλακες, ε, κάποια κενά που, που μπορεί να υπάρξει οικονομική δραστηριότητα στην εκάστοτε περιοχή και να καλύψει αυτό το κενό και να έχει έτσι συγκριτικό ε, πλεονέκτημα. Περιμένουμε ότι η ζήτηση για διάφορα μέταλλα θα αυξηθεί. Μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες σε αυτές τις περιοχές που ε, ε, στο παρελθόν ε, είχαν παραγωγή ενέργειας με υψηλή ένταση άνθρακα. Στη Γερμανία είδαμε ότι υπάρχει και βιομηχανικός τουρισμός και έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία. Δηλαδή κάποια ορυχεία πρώην εξορυκτικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει τόποι τουριστικού προορισμού και δείχνουν ε, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Και πολλά έχουν τύχει προστασίας από την UNESCO. Δηλαδή και ο τουρισμός μπορεί να αξιοποιηθεί. Τώρα πρέπει να έχουμε πολιτικές για τις δεξιότητες και τα προσόντα. Ε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ε, σχέδια για να προβλέψουν τις ανάγκες και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν. Έχουμε όμως και τις ε, βασικές τάσεις που επικρατούν τόσο ή άλλως τους η στην κοινωνια οπως ειναι η γυρανση του πληθυσμού και η ψηφιοποίηση. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να έχουμε ενεργές πολιτικές ε, στην αγορά εργασίας. Τι εννοούμε με αυτό. Να έχουμε πολιτικές ενεργητικές, να βοηθηθεί ο άναρχος να βρει δουλειά, είτε να αναπτύξει τα προσόντα του, τις δεξιότητές τους, είτε να ε, ταιριάξουμε καλύτερα με μηχανισμούς που έχουμε, θα έχουμε προβλέψει τα προσόντα και τις δεξιότητές τους με τα κενά στην αγορά εργασίας, με τις κενές θέσεις. το να μάθει κανείς πώς θα συγγράφει ένα βιογραφικό σημείωμα, το να μάθει πού θα ψάχνει για το κατά πόσο υπάρχουν και θέσει θέσεις και σε ποιο κλάδο της οικονομίας. Και αυτές τις, οι δεξιότητες αναζήτησης είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να καλλιεργηθούν. Το να προσπαθεί να ξαναμπεί κανείς στην αγορά εργασίας μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και πρέπει να μάθει πώς θα το κάνει. οι εργαζόμενοι από κλάδους υψηλής εντάσεις άνθρακα έχουν δεξιότητες που ταιριάζουν ε, και σε άλλους κλάδους που έχουν να κάνουν με την πράσινη ενέργεια και την πράσινη οικονομία. Πολύ συχνά δεν χρειάζεται να μάθουν και πολλά καινούργια ή πολλά διαφορετικά πράγματα και πρέπει να έχουν και εκπαίδευση στο επιχειρήν. Να ε, διδάξουμε στους ε, εργαζομένους, τους εκτοπισμένους πώς μπορούν να γίνουν αυτά απασχολούμενοι Πολύ συχνά το ποσοστό επιτυχίας ήταν σημαντικό, αλλά να σπρώχνουμε και να πιέζουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν τα προσόντα και δεν έχουν και την επιθυμία να είναι αυτοαποσχολούμενοι επιχειρηματίες, να τους πιέζουμε να γίνουν τέτοιοι, αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικές ε, ψυχολογικές συνέπειες αλλά και οικονομικές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι οι διαρθρωτικές πολιτικές. Η μετάβαση έχει να κάνει και την, ε, με την ανακατάσταση κατανομή του παραγωγικού input, δηλαδή των εργαζομένων, σε διάφορους κλάδους. Πρέπει οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες οικονομικές ευκαιρίες και πρέπει να θετήσουμε κατάλληλες πολιτικές. Πιο εύκολη διαδικασία να ξεκινήσει κανείς μια επιχείρηση, να παίρνει λιγότερο χρόνο, να συμμετάσχει ευκολότερα σε τέτοιου είδους προγράμματα, προγράμματα να έχουμε startup με χαμηλή ένταση άνθρακα. θα έχουμε μεγαλύτερες επενδύσεις, ανατομία και παραγωγικότητα, εάν επενδύσουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Πολλές πολιτικές δηλαδή πρέπει να εφαρμοστούν και απαιτείται χρηματοδότηση. Οι προηγούμενες εμπειρίες μας έδειξαν ότι πάρα πολλά κονδύλια δόθηκαν για να βοηθηθούν περιοχές να ολοκληρώσουν αυτή τη μετάβαση. Σήμερα όμως με τη δίκαιη μετάβαση και με τη μετάβαση σε χαμηλή ένταση ανθρακά τα πράγματα είναι πιο απλά. Έχουμε τον ενεργειακό φόρο ο οποίος ε, προσφέρει πολλά εισοδήματα στη χώρα. Όταν μιλούμε για 30 δολάρια ανά τόνο, χαμηλότερο από αυτό που έχουμε συζητήσει δηλαδή, αυτό στις χώρες του G20 θα οδηγήσει σε αύξηση 1% του ΑΕΠ. Δηλαδή, τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν σε κατά ποσό το οποίο θα είναι ίσο με αύξηση 1% του ΑΕΠ της εκάστοτε χώρας, της συγκεκριμένη χώρας. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά και είναι πηγή πόρων. Συνοπτικά λοιπόν και συμπερασματικά. Όπως δείχνουν οι προηγούμενες εμπειρίες αναδιάρθρωσης, χρειάζεται μία σειρά εργαλείων πολιτικής για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να ανακατεναμηθούν σε διάφορους άλλους κλάδες της ε, οικονομίας. Η μετάβαση χαρακτηρίζεται από δύο διαστάσεις φύλου που σχετίζονται μεταξύ τους και ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι υπερεκπροσωπούνται οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι στους κλάδους υψηλής έντασης άνθρακα ε, και ο αντίκτυπος της μετάβασης θα έχει πολύ μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπότα. Θα πάμε τώρα στον τρίτο εμπειρογνώμονα, τον κύριο Γκρέγκορη Πέις, από το Γραφείο Μελετών Μπρούγκελ ο οποίος θα αξιολογήσει την νομοπαρασκευαστική, νομοθετική μάλλον πρόταση, η οποία αξιολόγηση βεβαίως δεσμεύει μόνο εσάς και το ε, Ίδρυμα Μελετών σας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα το γυρίσω αμέσω στα αγγλικά, γιατί η παρουσίαση αυτή έγινε στα αγγλικά, ετοιμάστηκε στα αγγλικά σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την πρόταση αυτή και την ευκαιρία που μου δίνει να αξιολογήσουμε αυτή την σημαντική πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Βασικά στην εργασία αυτή που κάναμε, πραγματοποίησαμε μαζί με τρεις άλλους συναδέλφους από την Μπρούγκελ, προσπαθήσαμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που κάνουμε είναι να σας επισημάνουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία της πρότασης και το δεύτερο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια συνεκτική αξιολόγηση της πρότασης με, προτείνοντας και κάποιες πιθανές βελτιώσεις. Θα ήθελα να αρχίσω αμέσως τονίζοντας τα βασικά σημεία της πρότασης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί ακούσαμε πολύ λεπτομερή και πολύ ωραία παρουσίαση από την Κομισιόν. Θα σας συνοψίσω όμως τους βασικούς στόχους του νέου Ταμείου. Ε, ο δηλωμένος στόχος του Ταμείου, όπως βλέπετε εδώ, είναι να απαλύνει τον αντίκτυπο της μετάβασης, χρηματοδοτώντας τη διαφοροποίηση για τον εξυγχρονισμό της τοπικής οικονομίας και μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει. Στην πράξη σημαίνει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης βασικά θα δίνει επιχορηγήσεις για να χρηματοδοτηθούν τριών ειδών δράσεις βασικά που είναι η κοινωνική στήριξη, η υποστήριξη δηλαδή, του ανθρώπινου κεφαλαίου, η ε, οικονομική αναζωογόνηση προς τις επιχειρήσεις βασικά και αποκατάσταση της γης. Αυτά είναι τα τρία είδη δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν με αυτό το ταμείο. Όσον αφορά το μέγεθος του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα, η Κομισιόν προβλέπει ότι το Ταμείο θα βασίζεται σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ φρέσκο χρήμα, όπως λέγεται, από τον προϋπολογισμό του, ε, ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται θα προσθεθούν τα χρήματα αυτά στην πρόταση της Κομισιόν του 2018 για το MFF σε αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια θα προσθεθούν υποχρεωτικές μεταφορές από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ-ΣΥΝ ε, που έχουν δοθεί στα κράτη-μέλη ε, με ε, κρατική συγχρηματοδότηση και έτσι η συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων θα είναι γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε προηγουμένως η συνάδελφός μας από την Κομισιόν. Για το γεωγραφικό πεδίο, ε, το Ταμείο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά θα γίνει μια προκατανομή των κονδυλίων, η οποία θα βασίζεται σε μια αρκετά πολύπλοκη φόρμουλα, που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε δύο σημαντικά κριτήρια. Πρώτον, το ποσοστό εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου σε περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα, NATS ε, ε, S2, για όσους δεν το ξέρουν, οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν στις παλιές 22 περιφέρειες για τους Ισπανούς είναι η περιοχή, δεν ξέρω πώς λέγεται στα αγγλικά, είναι η αυτόνομες ε, περιφέρειες όπως λέγονται στην ε, Ισπανία. Αυτές είναι οι περιοχές ΝΑΤΣ 2 ε, και βασικά θα αναφέρεται αυτό το ποσοστό, καθώς επίσης και το ποσοστό των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα στην εξόριξη άνθρακα και λιγνίτη και στην σχετική βιομηχανία, σε τύρφη και σε σχιστόλιθο τι δράσεις θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Αναφέρονται 11 ε, τέτοιε δραστηριότητε που μπορούν να ομοδοποιηθούν σε τρει κατηγορίε, όπω ανέφερα προηγουμένω: κοινωνική στήριξη, οικονομική αναζωογόνηση και αποκατάσταση τη γη. Αναγέννηση των ε, ε, μολυσμένων περιοχών. Ε, Ακούσαμε ότι θα βασιστεί το όλο σύστημα στα εδαφικά σχέδια δίκαιη μετάβασης, όπου τα κράτη-μέλη θα εξηγούν πώς ε, προβλέπουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα στις ε, αντίστοιχες περιοχές και θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο τρόπο που θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα ε, θα είναι συμβατός με το στόχο τη ε, κλιματικής ουδετερότητας στο επίπεδο του κράτους μέλους. Και θα πρέπει τα σχέδια αυτά να εγκριθούν από την Κομισιόν για να ξεκλειδώσει η χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Θα ήθελα τώρα να έλθω στην ε, δική μας αξιολόγηση της πρότασης και να σας πω που βλέπουμε να υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης στον κανονισμό και που νομίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του η αξιολόγησή μας είναι αρκετά κριτική ή επικριτική αν θέλετε απέναντι στην πρόταση αυτή. Δεν είναι καλοπιστικού χαρακτήρα η προτάση μας, είναι ουσιώδης γιατί ε, θεωρούμε ότι έτσι το Ταμείο αυτό δίκαιη μετάβαση μπορεί να είναι χρήσιμο για τους πολίτες στη φάση της μετάβασης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η προέλευση του Ταμείου. Ε, θεωρούμε ότι είναι αφελές να θεωρήσει κανείς ότι αυτά τα ε, χρήματα που θα δοθούν στο Ταμείο θα είναι φρέσκο χρήμα πραγματικά ε, επιπλέον του MFF. Διότι ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το πολιετές πλαίσιο, ε, αλλά ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ των κρατών και του Κοινοβουλίου. Το ποσό αυτό του Ταμείου Δικής Μετάβασης θα ενταχθεί σε αυτό το ποσό που θα συμφωνηθεί. Άρα ε, το κατά πόσον αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια είναι φρέσκο χρήμα ή όχι ε, δεν έχει νόημα γιατί ξέρουμε ότι η διαφορά ε, ανάμεσα στις προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, άρα τα 7 εκατομμύρια δεν μετράνε πραγματικά, δισεκατομμύρια. Ε, επιπλέον, δεδομένου ότι ε, το ποσό αυτό θα ανήκει σε αυτό το συνολικότερο ποσό, ε, το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια θα αφαιρεθούν από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια. Κατά πάσα πιθανότητα θα προέλθουν από την πολιτική συνοχή, που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα χρήματα της δίκαιης μετάβασης θα είναι απλώς μια μετατόπιση των κονδυλίων συνοχής, δηλαδή 7,5 δισεκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τις πολιτικές συνοχή από κάποιες χώρες, και έχουμε εδώ μια εκτίμηση στην εργασία μας για το από πού θα φύγουν αυτά τα χρήματα και πού θα πάνε. Θα ε, φύγουν λοιπόν από κάποιες χώρες που τις βλέπετε εδώ, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ουγγαρία, ε, και θα δοθούν σε άλλες χώρες που είναι η Πολωνία, Γερμανία, ε, Τσεχία και Βουλγαρία βασικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο λοιπόν που πρέπει να σημειώσουμε. Και το άλλο είναι ότι είναι σημαντικό να ελέγξει κανείς ποια προγράμματα θα περικοπούν. Γιατί αν τα προγράμματα αυτά ε, είναι πολύ παρόμοια με τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Δικής Μετάβασης, τελικά ε, το Ταμείο αυτό δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια μετονομασία των πολιτικών χωρίς ε, κανένα πραγματικό διαφορετικό αποτέλεσμα. Τώρα, για το μέγεθος του ε, ταμείου και τους στόχους του, καταρχάς είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν προσπαθεί καν να αιτιολογήσει το ποσό αυτό σε σχέση με τους ε, στόχους και το πεδίο εφαρμογής. Τα αυτά τα 7,5 δις δεν ξέρουμε από πού κατέβηκαν και πώς βρέθηκαν σε αυτή την πρόταση. Το δεύτερο, επίσης είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια μέτρηση, ένα ποσοτικό υπολογισμό, αλλά η ανάλυση μας μας δείχνει ότι αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια θα είναι εντελώς ανεπαρκή για να καλυφθούν οι τρεις λειτουργίες που αναφέρθηκαν, η δηλαδή κοινωνική στήριξη, αναζωγόνηση της οικονομίας και αποκατάσταση της γης ε, δείχνουμε στην εργασία μας ότι μόνο η υποστήριξη των εργαζόμενων που θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω της μετάβασης θα απορροφήσει ολόκληρο αυτό το ποσό που πρόκειται να ανατεθεί στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Άρα κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να καλύψει και, τις τρεις, ε, αυτές, ε, και τους τρεις αυτούς στόχους που έχει θέσει το Ταμείο. Και γι' αυτό ε, έχουμε μία σύσταση στην εργασία μας που είναι να επανέλθουμε στην αρχική ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εστιάσει το Ταμείο αυτό μόνο στην κοινωνική υποστήριξη και σε ένα μικρότερο βαθμό στην αποκατάσταση της γης. Ξέρουμε ότι είναι κάπως ε, υπερβολική αυτή η πρόταση να γίνεται στην Επιτροπή Ρέτζι, αλλά κατά τη γνώμη μας δεν έχει νόημα να καταμεριστούν τόσο πολύ αυτά τα ποσά λόγω του μεγέθους των προκλήσεων και να διασκορπιστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε και πολλές και διάφορες δράσεις. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να εστιάζουμε την προσπάθεια σε μία βασική αποστολή που είναι η στήριξη της κοινωνίας, η κοινωνική στήριξη. Επίσης, η ανάλυση του καταλόγου των επιλέξιμων ε, δράσεων μας δείχνει ότι υπάρχει σαφώς επικάλυψη με άλλα προγράμματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι όλες οι δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα άλλα ε, ταμεία και από τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, χωρί να είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα εδαφικά σχέδια δίκαιη μετάβαση. Άρα, οι κύριε συστάσει μα είναι οι εξή. Πρώτον, Δεδομένου ότι προτείνουμε να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής, ε, θεωρούμε ότι ο κατάλογος των ε, επιλέξιμων δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιοριστεί ώστε να αντιστοιχεί στο μικρότερο αυτό πεδίο εφαρμογής να είναι οι επιλέξιμες δραστηριότητες αυτές που ε, έχουν τα γράμματα H, I, J και F στην ε, πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή βασικά νέες δεξιότητες και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, υποστήριξη αυτών που χάνουν τη δουλειά τους και αποκατάσταση της γης. Αυτή είναι η πρώτη μας σύσταση. Η δεύτερη σύσταση που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό ε, με αυτά που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος από τον ΟΣΑ, ε, πρέπει οι δραστηριότητε να είναι τέτοιε ώστε να γίνει η κοινωνική υποστήριξη πιο αποτελεσματική. Και εδώ πραγματικά θα πρέπει να ακούσουμε τον ΩΣΑ επί του θέματος αυτού για το upskilling και το reskilling και πώς μπορεί αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό, δηλαδή νέες δεξιότητες και αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Κάτι που αναφέρουμε στην ε, εργασία μας επίσης είναι ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατάρτιση ε, την εργασιακή και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Ε, καθώς επίσης και στην καταγραφή των νέων αναγκών. Διότι δεν έχει νόημα να πούμε θα κάνουμε κατάρτιση νέες δεξιότητες αν δεν ξέρουμε τι νέες δεξιότητες θα χρειάζονται. Επίσης κάτι άλλο που αναφέρεται και στην εργασία του ΩΣΑ είναι να συμπεριληφθεί κάποιο είδο ε, υποστήριξη του εισοδήματο αυτών των εργαζομένων. Γιατί όπω αναφέρθηκε ήδη λόγω του ότι κάποιοι από αυτού είναι μεγάλη ηλικία, ίσω ε, καλύτερο θα ήταν να του δοθούν κάποια επιδόματα που θα συμπληρώνουν τη σύνταξή του και ε, είναι σημαντικό, επειδή δεν ξέρουμε πού θα δημιουργηθούν καινούργιε θέσει εργασίας, να υπάρχει κάποια διευκόλυνση για την κοινωνικότητα. Ε, τέτοιου είδου δραστηριότητε και τέτοιου είδου δράσει θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση. Τέλο, επειδή συμπεριλάβαμε στι προτάσει μα και την αποκατάσταση τη γη, και για να γίνει σεβαστή η αρχή ο πληρώνει, η αποκατάσταση τη γη και η υποστήριξη για αυτήν θα πρέπει να περιοριζεται σε περιοχές όπου δεν έχει απομείνει καμία εταιρεία για να αναλάβει την αποκατάσταση, καμία επιχείρηση. Διαφορετικά θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, ε, το ότι λέμε ότι το Ταμείο θα πρέπει να εστιάζεται ε, στην ε, υποστήριξη την κοινωνική. Δεν θεωρούμε ότι η αναζωγόνηση της οικονομίας, δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι η αναζωγόνηση της οικονομίας δεν είναι σημαντική, είναι κρίσιμη σημασία, αλλά δεν είναι το Ταμείο Δικής Μετάβασης το καλύτερο εργαλείο για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άλλα εργαλεία, υπάρχει ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, ε, υπάρχει το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, αλλά και εκτός του προπολογισμού ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η δυνατότητα νέων επενδύσεων. Τέλος, όσον αφορά τη το γεωγραφικό καταμερισμό, θεωρούμε ότι αυτή η προκατανομή πολιτικά είναι κατανοητή για να πιστούν τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν με αυτούς τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους. Παρ' όλα αυτά ε, θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι οι πιο ε, άμεσα πληττόμενοι θα υποφεληθούν. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλύτερο να μην υπάρχει εκ των προτέρων ε, καταμερισμός και να ε, χρησιμοποιηθεί ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην... να χρησιμοποιηθεί μάλλον το μοντέλο που χρησιμοποιείται και για την, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, όπου τα ε, χρήματα δίνονται εκεί που υπάρχει η ανάγκη. Επίση, πέρα της, ε, του αν θα πρέπει να υπάρχει το προτέρων καταμερισμό, μα ανισχύει και η φόρμουλα που χρησιμοποιείται για τον καταμερισμό αυτό. Γιατί αν βάλουμε αυτά τα κριτήρια, ε, θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το χρησιμοποιεί τα επίπεδα όχι το, του ΝΑΤΣ 2, αλλά του ΝΑΤΣ 3. Ε, δείχνουμε στην εργασία μας ότι βασικά 40% των εδαφών του ΝΑΤΣ 3 που θα έπρεπε να αποφεληθούν από αυτό το ταμείο δεν ανήκουν στις ε, περιοχές ΝΑΤΣ 2 που μπαίνουν μέσα στον τρόπο υπολογισμού. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο τρόπος υπολογισμού δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις περιοχές που χρειάζονται τη βοήθεια αυτού του ταμείου. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό. Όσον αφορά τις συστάσεις, όπως έλεγα, θα προτιμούσαμε να μην γίνει καμία εκ των προτέρων κατανομή και να έχουμε ε, ένα μηχανισμό ανάλογο του EGF και αν γίνει εκ των προτέρων κατανομή, ε, γίνει δεκτή αυτή η μέθοδος, τουλάχιστον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, δεδομένα τον ε, του, του ΝΑΤΣ 3 ε, για να γίνει ο καταμερισμός αυτός, ε, ούτως ώστε να καλυφθούν οι σωστές περιοχές. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω, ελπίζω να μην μακρηγόρησα πολύ, ότι σχετικά με τις μεταφορές από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ Plus ε, στο Ταμείο Δικής Μετάβασης και σχετικά με την ιδέα αυτή ε, μεταφοράς από τα ΜΕΝ στο ΔΕ, το Ταμείο Δίκαιης Μετάφασης εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για κοινωνική στήριξη. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι λογικό να μεταφερθούν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δεν είναι καλό να συγχωνευτούν ε, οι δύο αυτές χρηματοδοτήσεις γιατί μια χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ε, το ένα ταμείο ή το άλλο ε, για να κάνει μόνο ε, κοινωνική υποστήριξη και, ή μόνο οικονομική αναζωγόνηση. Εμείς όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν και τα δύο ε, για να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι και οι δύο αυτές πολιτικές θα υλοποιούνται ταυτόχρονα σε κάθε δεδομένη περιοχή. Λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει ε, μεταφορά από το ΕΠΤΑ ε, στο Ταμείο Μετάβασης. Όμως, για να είμαστε βέβαιοι ότι και οι δύο αυτές προσπάθειες θα γίνουν ταυτόχρονα στο ίδιο περιφερειακό επίπεδο, καλό θα ήταν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν ένα τμήμα τουλάχιστον των, ε, του ΕΤΠΑ ε, στην οικονομική αναζωογόνηση των περιοχών που πλήττονται από την μετάβαση και που ε, θα εντοπίζονται με τα κριτήρια του Ταμείου Μετάβασης σαν ένα συμπλήρωμα προς την οικονομική, κοινωνική υποστήριξη που θα δώσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ξεπέρασα το χρόνο μου κατά δύο λεπτά. Αυτές είναι όλες οι συστάσεις μας όμως. Σας παρακαλώ ρίξτε μια ματιά και στην έκθεσή μας που είναι πολύ πιο λεπτομερής και αν έχετε ερωτήσει. σας παρακαλώ να μου τι θέσετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με email αργότερα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν ήξερα Προ τα που θα όδευαν οι συστάσει. Αλλά οι συστάσεις σας, όπως είπα και ευτυχώς που το είπα, δεσμεύουν μόνο εσάς. Και είμαι και βέβαιος ότι θα γίνουν πολλά σχόλια μεταξύ των συναδέλφων. Διότι μιλήσατε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Τουλάχιστον κάποιες από τις παρατηρήσεις σας ήταν πολύ ειλικρινής. Τώρα θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την προσέγγιση του εισηγητού μας, ε, του συναδέλφου μας Μανώλη Κεφαλογιάννη. Μανώλη, έχεις το λόγο. Thank you, President. I will be brief. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καταρχά θέλω να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ για τι ε, παρουσιάσει του στην Κομισιόν που μα παρουσίασε πολύ αναλυτικά την νομοθετική πρόταση. Να ευχαριστήσω όμω και ε, του εμπειρογνώμονε που μα παρουσίασαν στι διαφορετικέ πτυχέ του ζητήματο, διότι μα βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα και μας δίνουν και τροφή προσκέψη και συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Είναι μια προτεραιότητα επαριθμών 1 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να σας πενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το στόχο αυτό στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 η πρόταση για ένα ταμείο δίκαιης ε, μετάβασης. Είναι μια πρώτη νομοθετική πρόταση που εφαρμόζει την εν λόγω προτεραιότητα. Με τιμά ιδιαίτερα λοιπόν ε, και με καθιστά περήφανο ο ε, ορισμός μου ως εισηγητού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που είναι ένα πρώτο εργαλείο πολύ βασικό που θα εξασφαλίσει τη μετάβαση προς ε, μια οικονομία ουδέτερος προς το κλίμα με έναν ε, τρόπο δίκαιο που δεν θα αφήνει πίσω κανέναν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή. Κατά την άποψή μου όμως απαιτεί κάποιες ε, βελτιώσεις τις οποίες τη σημείωνα ε, και σίγουρα θα λάβω υπόψη ε, τις απόψεις των σκιωδών, άλλων ενδιαφερομένων συναδρέφων αλλά και τους που συμμετέχοντες στο όλο project. Όπως ε, γνωρίζετε, το Ταμείο Δικής Μετάβασης θα εδράζεται σε φρέσκο χρήμα της τάξης των 7,5 δις που θα δια... χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Και όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν πρόσβαση θα περιλαμβάνει ορισμένες μορφές επενδύσεων σε στοχευμένες περιφέρειες ανταποκρινόμενο στις διαφορετικές προκλήσεις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές κτλ. Αν θέλουμε να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δει ένα πολύ ευρύ φάσμα ζητημάτων και θα πρέπει επίσης ως κανονισμός να είναι ως το δυνατόν πιο ευέλικτος και στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του. Σε ό,τι αφορά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τον Ιούλιο ίσως να έχουμε την πρώτη θέση ανάως πριν από τις θερινές διακοπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα η σημερινή συζήτηση που κάνουμε θα πρέπει να ασχοληθεί με την προπαρασκευή της έκθεσης του σχεδίου έκθεσης των δυνατών και δεύτερον να θέσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πεδίο αρμοδιοτήτων διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μέχρι στιγμή, σε σχέση με το τελευταίο, οι επιτροπέ Μπάτ και Ίντ έχουν ζητήσει να είναι συναρμόδιες, καθήλων αρμόδιες και αυτές. Οι ΕΝΒΙ και η ΕΚΟΝ θέλουν να είναι συνδεδεμένες επιτροπές για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Η ΤΡΑΝ και η ΕΜΠΛ Περιμένουμε να θελήσουν να καταθέσουν γνωμοδοτήσεις. Ίσως χρειαστεί ένας μήνας μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Εμείς το μεταξύ όμως ήδη εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Τον Απρίλιο θα έχουμε τις τροπολογίες και το Μάη θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας την έκθεση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένος πως το μέλλον της Πράσινης Συμφωνίας ε, είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Έχουμε τα εργαλεία ε, για να το πετύχουμε και πιστεύω πως οι αρχές της δίκαιης μετάβασης ε, θα πρέπει να είναι πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι απλά ένα βήμα σε μια μακρά πορεία ώστε αυτή η προτεραιότητα να λάβει σάρκα και ωστά. Εγώ προσωπικά θα είμαι επικοδομητικό, θετικά διακείμενο, διαθέσιμο σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή για να συζητήσουμε τι ιδέε, ανησυχίε, προτάσει τις προτεραιότητές τους. Ε, και φυσικά θα συνεργαστώ στενά και με τους σκιώδεις εισηγητές, τους συμβούλους, ε, συνεργάτες, τα κράτη-μέλη και τις ε, διγόμενες περιφέρειες. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας και τη συνεισφορά σας στο το Κοινοβούλιο να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα και να έχουμε έναν καλό κανονισμό εγκαίρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την υποστήριξη και την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε βέβαιος, να είστε βέβαιος ότι θα έχετε την υποστήριξη όλου του προσωπικού της Επιτροπής Ρέτζι για το έργο που ξεκινάτε. Απλά θέλω να προσθέσω πως υπάρχουν προφανώς και κάποια ερωτηματικά από την πλευρά του Συμβουλίου, διότι είμαστε σε στάση αναμονής. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Και για τα δημοσιονομικά περιμένουμε και για το χρονοδιάγραμμα περιμένουμε. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πέντρο Μάρκες για μια πρώτη παρέμβαση, εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Από την πλευρά των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα θέλαμε καταρχάς να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει κατά την άποψή μας ε, αυτό το εργαλείο. Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ε, και να προωθήσουμε την οικολογική, την πράσινη μετάβαση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και τις επιπτώσεις που θα έχει και το κοινωνικό σύμφωνο. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι ένα ενδεδειγμένο εργαλείο αυτό. Υπάρχουν ωστόσο προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο έργο αυτό που ξεκινούμε. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο, τους συντονιστές, για το πολύ ποιοτικό αυτό εργαστήριο. Ακούσαμε ποιοτικέ παρεμβάσεις, ακούσαμε θαραλές προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη του εισηγητή και σκιώδη εισηγητέ, αλλά και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο εν Άκουσα με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή ε, γιατί μίλησε έτσι με πολύ θάρρος ε, για τη δουλειά αυτή που μόλις ε, ξεκινά. Θέλω να επιμείνω στην κοινωνική διάσταση της μετάβασης. Ακούσαμε προτάσεις συστάσεων που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η πράσινη μετάβαση, και το έχουμε πει και στη δική μας πολιτική ομάδα, θα πρέπει να έχει και μία, αν μπορώ να το πω έτσι, κόκκινη πτυχή. Καλή πράσινη μετάβαση, όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ταυτόχρονα την ψηφιοποίηση και την ε, απαλλαγή, την εγκατάλειψη του άνθρακα. Επομένως, αυτή η πράσινη ε, συμφωνία ε, είναι ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην κοινωνική διάσταση εκμεταλλευόμενοι τους άλλους πυλώνες του μηχανισμού δικές μετάβασης ιδίω ό,τι αφορά την οικονομική μετάβαση. Δεν έχουμε πολλά μέσα, δεν έχουμε πολλού πόρου στη διάθεσή μα. Επομένω, θα πρέπει να στηρίξουμε τα εδάφη μα, τι περιοχέ και του ανθρώπου που ζουν ε, πολύ κοντά στη μετάβαση. Ως ε, διαχειριστής ε, δημόσιων πολιτικών έχω διαπιστώσει ότι σε πολλά από τα εδάφη που θίγονται από, και έχουν θίγει κατά το παρελθόν από ε, τις βιομηχανικές εξελίξεις υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι θα βρουν μια άλλη δουλειά και με ένα μαγικό ραβδάκι θα αλλάξουν δεξιότητες και θα βρουν τη θέση τους και μια δουλειά στη νέα οικονομία. Υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού για τις περιφέρειες αυτές και για πολύ κόσμο. Στις περιφέρειες, λοιπόν, στα εδάφη ε, τα οποία θα θυγούν, Υπάρχουν και κάποιες περιοχές ε, που αντιμετωπίζουν περισσότερο κίνδυνο και έχουν ήδη κατά το παρελθόν ε, αντιμετωπίσει προβλήματα, έχουν πληγεί από τη βιομηχανική μετάβαση εγκατέλειψαν ε, τη βαριά βιομηχανία. Ήδη λοιπόν είναι εδάφη που βρίσκονται σε υποβάθμιση, σε παρακμή. Και πρέπει να τις βοηθήσουμε, τις περιφέρειες πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, ισχυρή βιομηχανική βάση στις περιφέρειες αυτές ε, που θα ε, πλαισιώσει την πράσινη μετάβαση. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ώστε να διατηρηθεί η απασχόληση να διατηρηθούν θέσει εργασία. Άρα πρέπει να δουλέψουν πάνω στην κοινωνική διάσταση. Πολλοί εργαζόμενοι σίγουρα μπορούν, αν τους δοθεί απαραίτητη βοήθεια, να μεταβούν σε μια νέα ε, φάση της ζωής τους. Ασχολούμαι, παραδείγματος χάρη, με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, ε, με κοινωνικές υπηρεσίες, ε, κοινοφελείς υπηρεσίες μπορούν να δημιουργηθούν θέσει εργασίας. Όπως είπε όμω και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, αυτή η μετάβαση και αυτά τα μέσα εργαλεία υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών θα μείνουν στα λόγια, στα ωραία λόγια, εάν δεν συνοδευτούν από επαρκή φιλόδοξη χρηματοδότηση, φιλόδοξο προπολογισμό. Οι προτάσεις ε, του Προέδρου Σάρλ Μισελ μας φαίνονται πολύ καλές, διότι έρχονται να προσθεθούν στο Τάμιο Δικές Μετάβασης ε, και το έχουμε πει ομόφωνα εμείς ως Κοινοβούλιο ότι είμαστε κατά της πρότασης εμβάσματος μεταφοράς πιστώσεων γιατί αν θέλουμε ε, να πιστέψουμε ότι είναι φρέσκο αυτό το χρήμα, νοπό, από κάπου πρέπει να βγει. Δηλαδή να δώσει 1% το κάθε κράτο μέλο και να έχει ίσχυτη τη σύνδεσή του. Όχι. Αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει ένα μοχλό ευρωπαϊκή πολιτική, χρειάζεται και επαρκή χρηματοδότηση. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα ε, κονδύλια, περισσότερο νοπό χρήμα και όχι μεταφορά πιστώσεων. Και κάτι τελευταίο. Πρόκειται για μια μετάβαση που θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει καιρό και πρέπει να ληφθεί υπόψη και η έξω κοινοτική διάσταση. Τι γίνεται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιομηχανία μα, η κοινωνική συνοχή, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν θα μπορέσουν να ανθέξουν, δεν θα μπορέσουν να διαρκέσουν αν δεν μα απασχολήσει και το ζήτημα τη παραγωγή άνθρακα εκτό συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν εντάσσεται στο Ταμείο Δική Μετάβαση. Ωστόσο, περιλαμβάνεται στι γενικότερε φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είχα να πω εισαγωγικά και θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή του υπόλοιπου συναδέλφου. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Pedro. Ευχαριστώ πολύ τον Πέδρο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νοτέξ και ο δισηγητή και συντονιστή για το Ρινιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους προλαλήσαντες για τις πολύ επικοδομητικές τους παρουσιάσεις για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και για τις ανθρακοπαραγωγικές περιοχές που βρίσκονται σε φάση οικονομικής μετάβασης. Ε, χαιρόμαστε διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνένταξε την πρόταση πολύ γρήγορα. Ήταν μία από τις υποσχέσεις της Επιτρόπου Ελίζα Φερέιρα. Οι πολίτες ζητούν στήριξη και αυτό είναι πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε πρόταση αληθινή, επιτάπητο, στα χέρια μας και μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Αρχικά η ιδέα ήταν πια με αυτό το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση να αφορά μόνο τι ανθρακοπαραγωγικέ περιοχές. Είναι σαφές όμως τώρα πια ότι για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματική αλλαγή πρέπει να εμπλέξουμε εκεί περισσότερες περιφέρειες, να εντάξουμε περισσότερες περιφέρειες. Άρα θα πρέπει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης να συνοδεύεται και να πλαισιώνεται από μηχανισμό, από διευκόλυνση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες διαφόρων κλάδων και διαφόρων περιφερειών. Δύο είναι τα ερωτήματα που έχουμε βασικά να απευθύνουμε στους ομιλητές. Πρώτον, για το ύψος της χρηματοδότησης. Θα είναι αρκετά τα χρήματα. Εγείρονται ανησυχίες, εκατέρωθεν από πολλές πλευρές ότι η προτινόμενη χρηματοδότηση του Ταμείου για τη δίκαιη μετάβαση δεν θα είναι επαρκής, ούτε η χρηματοδότηση του JTM. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Αν αυτά τα εργαλεία θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, θα μπορέσουν να στηρίξουν όλες τις επενδυτικές ανάγκες. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας υπάρχουν περιφέρειες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά. Ορισμένες ανθρακοπαραγωγικές περιφέρειες. Ήδη το βλέπουμε να χάνονται θέσεις απασχόλησης ή θα χαθούν τους επόμενους μήνες. και πολλές, μάλιστα. Και ταυτοχρόνω κάποιες πόλεις σε αυτές τις περιφερείες αντιμετωπίζουν τον άμεσο κίνδυνο της ε, ε, διακοπής της κεντρικής θέρμανσης ε, και της παροχής νερού. Το είδα την Παρασκευή εγώ που πήγα σε αποστολή σε ανθρακοπαραγωγική περιοχή. Θα διακοπεί. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχης από αυτές τις περιφέρειες που έχουμε υψηλή ένταση άνθρακα επιδιώκουν λύσεις, επιζητούν λύσεις, αναζητούν επενδυτές. Στηρίζονται συχνά από τις εθνικές κυβερνήσεις σε κεντρικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, για να έρθει νέος επενδυτής θα έρθει στην περιφέρεια μόνο αν έχει διασφαλίσεις και εγγυήσει ότι θα βρει και εργαζομένους. Και οι απασχολούμενοι εργαζόμενοι, αν χάσουν τη δουλειά τους στα... στην ανθρακόβιομηχανία, θα μείνουν στην περιφέρεια μόνο αν τη βρουν ελκυστική. Ή αλλιώς θα φύγουν. Και τι σημαίνει να είναι ελκυστική η ζωή στην περιφέρεια. Να έχουν νοσοκομεία, να έχουν σχολεία, να έχουν δρόμου, βασικέ υποδομέ. Άρα βλέπετε ε, πόσες πολλές διαστάσεις περιλαμβάνει και περικλεί αυτό το ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση. Είναι ζωτική σημασία να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι κάτι που ξεπερνά το JTF, το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση και το μηχανισμό και τη διευκόλυνση για τη δίκαιη μετάβαση του JTF και του JTM δηλαδή αντίστοιχα. Έχει να κάνει όλο αυτό και με το, το πολιτική συνοχής όλα αυτά ε, είναι χρήσιμα. Θα είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο και επιτυχημένο, πιστεύουμε. Συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε για τον προπολογισμό που συνοδεύει το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι αρκετό ο προπολογισμό, αλλά ο χρόνο θα το δείξει αυτό. Οι πολίτε αξίζουν τη στήριξή μα. Και τέλο. Αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Θέλουμε συνεργασία μελλοντικά και σε τεχνικό επίπεδο για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβαση. Ευχα... Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο και εγώ σα ευχαριστώ, Αντρέη, για τους πράσινου Χίτλα Νίνας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε. Πρώτα, πρέπει να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ποιο είναι ο στόχος του Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση, προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε, πού θέλουμε να φτάσουμε. Πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Είναι ίσονο σημασία στο γεγονό ότι μια, ένα από τα ελάχιστα καλά Τη πρόταση ε, του Μισελ, του κυρίου Μισελ από το Συμβούλιο, είναι ότι για να πάρει κάποιο στήριξη πρέπει να έχει δεχτεί σταδιακά να εξαλείψει την άνθρακο παραγωγή. Είναι μια επίδειξη καλής θέλησης. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Το Ταμείο Δίκης Μετάβασης υπάρχει για να στηρίξει τον οποιονδήποτε θέλει να φύγει από τον άνθρακα και θέλει να λύσει αυτό το ζήτημα του περιβάλλοντος θα πρέπει λοιπόν να καταγραφεί επισήμως και όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού ότι είναι ένας χρυσός κανόνας και πρέπει να καταγραφεί στη συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση. Υπάρχει στην πρόταση της Κομισιόν και δεν θέλουμε να βγει αυτό, να αφαιρεθεί. Η μετάβαση προς τις πράσινες πηγές ενέργειας μπορεί να τύχει στήριξη για να στήριξεις για να ελευθερωθούμε πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Από εκεί και πέρα πολλά έχουν υποθεί. Μεγάλο είναι το πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Θέλαμε φρέσκα χρήμα και πιστεύω ότι τα 7,5 δις ευρώ δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά έργα που έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο οι υπολογισμοί αυτοί θα μεταφραστούν στην πράξη, έτσι όπως προτάθηκε στην αρχή. Ζητήσαμε, αναζητήσαμε συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία υπήρξε αυτό το αίτημα. Είναι επικίνδυνο να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να πάρει χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία καλύπτουν τόσο πολλές ανάγκες και να τα βάλει στις ίδιες περιφέρειες οι οποίες ε, παίρνουν χρηματοδότηση και από αυτά και από το Ταμείο Δικής Μετάβασης. Δηλαδή, ε, τι κάνουμε, παίρνουμε χρήματα από μια περιφέρεια έτσι και τα μεταφέρουμε στην άλλη περιφέρεια. Θα είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και αν δεν γίνει σωστά, στο τέλος θα πληγούν περισσότεροι, γιατί οι περιφέρειες που επωφελούνται από τα διερθρωτικά ταμεία θα χάσουν τη χρηματοδότηση, άρα οι άνθρωποι τους θα χάσουν χρηματοδότηση και ε, θα πληγούν ούτως ή οι άνθρωποι που είναι στις περιφέρειες που θα επωφεληθούν από το Ταμείο Δικής Μετάβασης ε, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Νομίζω ότι ο εισηγητής πρέπει να τα εξετάσει αυτά εξαιρετικά προσεκτικά και ε, ε, ε, να καλύψει με πολύ μεγάλη προσοχή αυτές τις λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, με αυτή τη διευκόλυνση, με αυτό το μηχανισμό και τη συγχρηματοδότηση και τι εγγυήσει και το καθεξής και όπως λέγονται τέλος πάντων, καλό είναι άμα δουλέψουν όλα αυτά, αλλά ε, για να σας μιλήσω ειλικρινώς, προτιμώ να έχω ένα σχέδιο που θα δουλέψει ε, ανεξαρτήτως εξελίξεων. Δηλαδή δεν με νοιάζει αν θα είμαστε σε έναν ενάρετο οικονομικό κύκλο και η οικονομία θα είναι σε καλή φάση. Θέλω ένα σχέδιο που θα δουλεύει και όταν η οικονομία πάει καλά και όταν δεν πάει. Χρειαζόμαστε μια, ένα σταθερό εργαλείο χρηματοδότησης έτσι ώστε να χρηματοδοτούμε αυτό το Ταμείο Δικής Μετάβασης όχι μόνο για την επόμενη 7 ετία, αλλά για την επόμενη 20 ετία. Και για να το πετύχουμε αυτό δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που λαμβάνουν χώρα κάθε 7 χρόνια. Προτιμώ χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, επιβιώσει και να μακροημερεύσει για τα επόμενα 20 χρόνια και να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους, να τους κοιτάξουμε κατάματα και να τους πούμε ορίστε η πηγή των χρημάτων για να κάνετε με μετάβαση με δίκαιο τρόπο τα επόμενα 20 χρόνια εσείς στις περιφέρειές σας. Τώρα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επανειλημμένως έχουμε πει ότι είναι όνειδος, είναι ντροπή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αυτό που προτείνει το Συμβούλιο, αυτό που προτείνει ο κύριος Μισελ διότι δεν ανταπεξέρχεται στα πρότυπα που έχουμε και στις προσδοκίες. Γιατί ζητούμε όλο και περισσότερη δουλειά να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τη χρηματοδοτούμε, χωρίς να της δίνουμε τα μέσα να τη φέρει σε πέρας. Ελπίζω να είμαστε σε θέση να πείσουμε τους πολιτικούς μας στις ε, χώρες μέλη να δώσουν περισσότερα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε να αγωνιστούμε για μεγάλους, για υψηλούς σκοπούς, για υψηλά ιδεώδη, για το ευρωπαϊκό μέλλον που είναι και το μόνο μέλλον σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Με χαρά θα συνεργαστώ με όλους σας και με εσάς ε, και τους εκπροσώπους από τα διορθωτικά ταμεία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ, Νίκολας. Αντρέι Νόβακοφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους αξιότιμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του JGRC και του μελετητικού γραφείου που έχει εκπονήσει αυτή την έρευνα του Ιδρύματος Μπρούκελ και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές για τη δουλειά τους. Πολλά ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν και εξηγήθηκαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων με επίκαιρο τρόπο και με άξιο τρόπο. Τονήθηκε λοιπόν το θέμα της ισότητας των φύλων στα ανθρακοριχεία. Ταπεινή μου συμβουλή είναι να μην βιαστούμε αυτά να τα κάνουμε πράξη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει δεκτή η ιδέα ε, με επεφημίες εν χορό από τις τοπικές μας κοινωνίες. Έρχεται το New Green Deal, η νέα πράσινη συμφωνία. Αυτό είναι βέβαιο. Ακόμα και αν δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, η νέα πράσινη συμφωνία είναι προ των πυλών. Άρα, πρότιμο ο εισηγητής, οι σκιώδες εισηγητές, ε, όλη η ομάδα Ρέτζι να είναι πιλότοι σε αυτό το τρένο, να είναι οδηγοί, καπετάνιοι και όχι επιβάτες μόνο. Άρα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως θεσμικό όργανο το οποίο έχει και την τελευταία λέξη να πει σε αυτή τη διαδικασία. Και όπως είπα και στην αρχή, σίγουρα όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα στηρίζουν τη νέα πράσινη συμφωνία. Όλοι θέλουν πιο καθαρό αέρα, πιο καθαρό νερό, πιο, πιο υγιεινό, πιο καθαρό φαγητό ε, στο τραπέζι για μας και την οικογένειά μας. Θέλουμε όμως να είμαστε πράσινοι και φτωχοί συνάμα. Ταυτοχρόνως δεν το πιστεύω. Κάθε ΜΒ το οποίο μετασχηματίζεται από πηγή άνθρακα σε πηγή ανανεώσιμης ενέργειας μεταφράζεται σε απώλεια θέσης απασχόλησης ε, για κάποιες περιφέρειες. Κάθε ΜΒ που χάνεται κατά τη διάρκεια αυτή του μετασχηματισμού του μπορεί να οδηγήσει σε στραγγαλισμό για την βιομηχανία μας. Στηρίζω τη Νέα Πράσινη Συμφωνία και θα συνεχίσω να τη στηρίζω με όλους τους τρόπους, όμως να γίνεται αυτή και να εφαρμόζεται σε βαθμό και με ρυθμό ε, με τον οποίο να μπορεί να προσαρμοστεί η οικονομία μας. Σίγουρα θα βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε με αυτό τον τρόπο, με έτσι, με αρμονία και με τους συναδέλφους που ε, θα συνεργαστούν για την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια έκθεση πολύ καλά ισορροπημένη και σε πολιτικό επίπεδο και σε γεωγραφικό επίπεδο και σε κάθε άλλο δυνατό επίπεδο. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή αρχή και αυτή η πολύ καλή αρχή θα μας οδηγήσει σε έκθεση σε ε, ε, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιμένοντας βεβαίως από το Συμβούλιο να αποφανθεί επίση από την πλευρά του. Καλό τους συναδέλφους να στηρίξουν τη Νέα Πράσινη Συμφωνία, το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση, αλλά να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε ακριβώς λόγω ε, του άνθρακα και του χάλιβα. Χάρη σε αυτά υπήρξε αρχικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σκιώδης εισηγητής συνάδελφος Ντονάτο ήταν παρόν, δεν τον βλέπω όμως. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους και την Κομισιόν που με τις ε, παρουσιάσεις τους μας βοήθησαν να ξεκινήσουμε αυτή την σημαντική συζήτηση ε, στην οποία είναι φανερό ότι για μας τουλάχιστον παραμένουν πολύ μεγάλες απορίες και ερωτηματικά που προέκυψαν και από την συζήτηση αυτή. Θα ξεκινήσω από τις δικές σας ε, σκέψεις, Πρόεδρε, στην αρχή που παρουσιάσατε ε, για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αυτό σχετίζεται άμεσα με το θέμα το οποίο συζητάμε. Η εργασία που πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου σε αυτή την Επιτροπή είναι μια εργασία πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι το πρώτο πραγματικό φίλτρο που μας επιτρέπει να μπούμε στην ουσία σε σχέση με τις πολλές και διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει στις τόσες πολλές συζητήσεις που έγιναν αυτούς τους μήνες από τότε που ε, ε, ανέλαβε καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να μπούμε στην ουσία, γιατί υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Η πρώτη αμφιβολία που προέκυψε σαφέστατα είναι ποια είναι η πραγματική οντότητα των κονδυλίων αυτών που θα χρηματοδοτήσουν αυτό το Ταμείο Μετάβασης. Αυτή η θεώρηση του φρέσκου χρήματος, όπως λέγεται αυτές τις μέρες, ε, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί και η συζήτηση που γίνεται για το MFF μας δείχνει ότι αν θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι ε, με τα τρία τραπουλόχρητα, να παίξουμε τον παπά, τελικά θα είναι σαν να παίρνουμε τα χρήματα αυτά ε, από κάπου αλλού και να τα φέρνουμε εδώ. Και ε, παίρνουμε από κάπου και βάζουμε κάπου αλλού. Ε, αυτό φαίνεται να γίνεται. Άρα οι αμφιβολίες για την προέλευση αυτών των κονδυλίων είναι προφανείς. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ανομαλίες όμως, ε, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε μεγάλη προσοχή. Η πρώτη από αυτές ε, αφορά τα ε, μια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Πρέπει να ε, καταλάβουμε αν πραγματικά μιλάμε για επιπλέον πόρους ή απλώς ε, φανταζόμαστε ένα μεγάλο ποσό στα πλαίσια αυτού του New Deal που είναι απλώς μετατόπιση, μεταφορά κονδυλίων. Εγώ βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την παρέμβαση του κυρίου Κλέιερς που έθεσε τα πιο κρίσιμα σημεία. Την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί τα θέματα που ε, ανέδειξε είναι θέματα που κάποιοι μας τα αναφέρουμε εδώ και πολύ καιρό, άλλοι που δεν το, τα αναφέρουν ρητά, αλλά είναι αντικειμενικά ε, στοιχεία και συνοδεύουν αυτές τις συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε αυτές τις πτυχές και πιο συγκεκριμένα τι επιπτώσεις θα έχει αυτό για την πολιτική συνοχής, ούτω ώστε να μην υπάρξουν χώρες οι οποίες θα επιβαρυνθούν δύο φορές από αυτή την επιλογή. Από τη μια μεριά με τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων και από την άλλη με τις περικοπές στην πολιτική συνοχής. Ενώ οι χώρες αυτές δεν θα ε, επωφεληθούν κατά ανάγκη από τα προγράμματα για τα οποία ε, μιλάμε. Αυτή μπορεί να είναι η πραγματικότητα. Έτσι πιστεύω λοιπόν ότι οι εργασίες που θα γίνουν ε, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε τα κριτήρια ε, στα οποία βασίζονται οι επιλογές αυτές. και για να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για τα μαθηματικά στοιχεία και την εκ των προτέρων ε, κατανομή των κονδυλίων δεν είναι κάτι ε, υποχρεωτικά, υποχρεωτικά θετικό αυτό πριν καταλάβουμε ποια είναι η ουσία του προγράμματος. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το θέμα των διορθώσεων που προτείνονται και που θα πρέπει να συζητηθούν επί τη ουσία και σε βάθο. Δεν θα πούμε βέβαια σε αυτή τη συζήτηση τώρα, να το αναφέρω σαν τίτλο. Ένα άλλο θέμα είναι το κριτήριο που αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν βιομηχανίες υψηλής ένταση άνθρακα στο επίπεδο ΝΑΤΣ 3. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν χρησιμοποιείται για παράδειγμα το κριτήριο ε, Eurostat. Όλα αυτά είναι σημεία ε, στα οποία αξίζει να εμβαθύνουμε και να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί, και θα κλείσω με αυτό, έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θέμα το οποίο ζητάμε σήμερα μα βρίσκει όλους σύμφωνους. Ακόμα και αν εγώ ε, δεν τοποθετήκα θετικά η ομάδα μου απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν. Δεν το κάναμε αυτό γιατί διαφωνούμε με το στόχο, αλλά διότι τους τελευταίους μήνες μας δημιουργήθηκαν κάποια μεγάλα ερωτηματικά που δυστυχώς ε, ακούσαμε να επιβεβαιώνονται σήμερα σε τεχνικό επίπεδο και θα πρέπει να βρουν απαντήσεις. Και η συζήτηση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί στην Επιτροπή μας αφού δοθούν οι απαντήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ΚΟΕ η Μαρτίνα Μισελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι θετικό το ότι η Κομισιόν μια από τις πρώτες της προτάσεις στο πλαίσιο της νέας πράσινης συμφωνίας κάνει αυτή την πρόταση για αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και αυτό σε σχέση και με το στόχο να ληφθεί υπόψη κοινωνική διάσταση, να ενισχυθεί δε η κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πω ότι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε ε, και σε άλλες διαδικασίες ε, ε συζήτησης ε, να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας να είμαστε συνοδηγοί, αλλά να έχουμε το νου μας πολύ καλά στο δρόμο που ακολουθούμε. Διότι ήδη υπάρχουν κάποια πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία τίθενται στο πλαίσιο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί επιτάπητος και μάλιστα ε, μας κάνουν να διαρωτώμαθα ακόμη περισσότερο ιδίως μετά από αυτά που ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του Μπρούγκελ και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά. Μιλάμε για νοπό χρήμα, ειλικρινά, όταν από τη μία πλευρά αυτά τα 7,5 δις θα πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά ε, με τις προτάσεις που ακούσαμε και έχουμε και την πρόταση του Συμβουλίου που ήδη διαγράφει κονδύλια από την ε, πολιτική συνοχής. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να μιλήσουμε για νοπό χρήμα, σε καμία περίπτωση. Επίσης είναι θετικό το ότι επί της αρχής τουλάχιστον ε, θα μπορεί, θα πρέπει να αποφεληθεί κάθε κράτος μέλος από αυτό το Ταμείο Μετάβασης. Υπάρχει όμως και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που δεσμεύει όλα τα κράτη. Γιατί λοιπόν τα μισά από αυτά τα χρήματα ε, δεν έχουν ε, σύνδεση με αυτόν το, στόχο. Και αν ε, έχουμε αυτά τα ποσά του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ που προτείνονται για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, εδώ μιλάμε ουσιαστικά για πρόσθετη περικοπή των κονδυλίων συνοχής που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η πολιτική συνοχής για την ίδια την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η χρηματοδότηση λοιπόν τελικά τι ακολουθεί. Ακολουθεί τις επιταγές ε, του Ταμείου Δίκαιης ε, Μετάβασης ε, ή του ΕΚΤ Plus, του ΕΚΤ ΣΥΝ. Τι θα γίνει με τη συγχρηματοδότηση. Και αυτό την, τον επιμερισμό ΝΑΤΣ 3. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ε, δυνατότητα επίσης ε, αναδιάρθρωσης ή ε, ανακύκλωση των εργαζομένων και τι θα γίνει και σε ε, περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε αυτά τα σχέδια που απλά ανακυκλώνονται ή λαμβάνονται υπόψη ε, οι νέες ενδείξεις και τα νέα στοιχεία και λαμβάνουμε υπόψη και το προσδόκιμο επιβίωσης και πολλά άλλα στοιχεία. Είναι ερωτήσεις όλες αυτές που προκύπτουν. Ο κύριος από τον Μπρούγκελ έκανε και κάποιες συστάσεις στο τέλος της παρέμβασής, της παρέμβασής του. Ας περιοριστούμε στη στοχοθέτηση αλλά κυρίως θα έλεγα στις κοινωνικές επιπτώσεις και στις απώλειες θέσεων εργασίας Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και νομίζω στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να τα θέσουμε με ειλικρίνεια. Δεν πάνε όλα, δεν περιστρέφονται όλα γύρω από το χρήμα, αλλά είναι θέμα στοχοθέτησης ε, και επιδιώξεων. Περιμένω να γίνει αυτός ο διάλογος, αυτή η κοινή συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μαρτίνα. Ερχόμαστε στο τέλος του πρώτου γύρου των συζητήσεων με τον εισηγητή και τους σκιώδη εισηγητές. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα παρόντα μέλη. Αν θέλετε όμως, α... ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή ε, για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης από την Επιτροπή των Περιφερειών, ο κύριος Ομπερζέη, που ε, μας θυμάμαι την παρουσία του και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας συστηθώ. Είμαι ο Βόι Ογκερσέλ, δήμαρχος της πόλης Ιέρικα, και εισηγητή για το Ταμείο δίκαιη μετάβαση εκ μέρου τη επιτροπή των Περιφερειών. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε εν συντομία την ευκαιρία να παρουσιάσω τα βασικά σημεία της γνωμοδότησής μου από την οπτική γωνία των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα κατά την συζήτηση αυτή που προηγήθηκε. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα συντάξει τη γνωμοδότησή της πολύ, σύντομα ε, και γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ θα έλεγα, γιατί περιμένουμε στις 25-26 Μαρτίου ε, φέτος να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Τα κύρια σημεία αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης είναι πολύ παρόμοια με αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής εδώ, Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν μπορεί να ε, αντικαταστήσει ε, περικοπές στην ε, πολιτική συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη τους όταν θα συζητούν το MFF. Περιμένουμε λοιπόν να, υπάρχει όντως νέο, να υπάρξει νέο χρήμα. Η οικονομική υποστήριξη πρέπει να συνδέεται με δέσμευση στους στόχους του Green Deal και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, σαφής δέσμευση με μια ε, ε δίκαιη ε, μετάβαση πραγματικά, ε, συμμόρφωση με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, ε, τον στόχο μας για το 2050 όσον αφορά τις περικοπές των εκπομπών και για τον στόχο για το 2030 σχετικά με την περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θερμοκηπίου, ανθρακούχων εκπομπών κλπ. Όσον αφορά τα εδάφη που θα υποφεληθούν, θα πρέπει να είναι οι περιοχές ή μάλλον με συγχωρείτε, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στις περιοχές ε, ΝΑΤΣ 3, θα πρέπει να εστιαστούμε στο επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Γιατί? Γιατί όλα τα διαρθρωτικά ταμεία εφαρμόζονται ε, στα επίπεδα ΝΑΤΣ 2 και αυτό σημαίνει ότι θα απλοποιηθεί έτσι η διακυβέρνηση του ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ε, προκειμένου να αποφασίσουν για τα ποσά που θα μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αντί να οριστεί το ποσοστό στη χρηματοδότηση σε ένα ελάχιστο μία μισή φορά ε, και σε ένα μέγιστο ε, τρεις φορές ε, το κονδύλι του Ταμείου, ε, θα πρέπει ε, το ελάχιστο είναι το μισό της χρηματοδότησης και το μέγιστο τριπλάσιο, από μισέως τριπλάσιο. Ε, επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει πολύ σαφές ότι οι δραστηριότητες που οδηγούν σε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να εξαιρούνται, να αποκλείονται από την ε, δυνατότητα χρηματοδότησης. Και τέλος θεωρούμε ότι η πλατφόρμα για τη δίκαιη μετάβαση που θέσπισε η Κομισιόν για να διευκολύνει την διμερή και πολυμερή ανταλλαγή ε, εμπειριών ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ετήσιο φόρουμ των περιοχών της δικής μετάβασης, ώστε να γίνεται εκεί μια πολιτική ανάλυση της πρόοδου που έχει γίνει σχετικά με τους στόχους του Ταμείου Δικής Μετάβασης και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ε, πρόθυμη ε, να αναλάβει ε, οργανωτικό ρόλο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώνει δηλαδή αυτό το ετήσιο φόρουμ της δικής μετάβασης. Δεν θα είναι εύκολο να υλοποιηθούν όλα αυτά, αλλά όλα τα ταξίδια, ακόμα και τα πιο μακρινά, ξεκινάνε με ένα πρώτο βήμα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Je veux informer notre... Ευχαριστώ να ενημερώσω τον εισηγητή μας πως ναι, βάλτε τα ακουστικά. Ε. Έλεγα λοιπόν, να σας, έλεγα, ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει και αυτή κάνει την εργασία της, το οικονομικό τμήμα συγκεκριμένα, η Οικονομική της Επιτροπή για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Οπότε στην πρώτη αυτή ε, ημερίδα ε, θα ακούσουμε και την ΕΟΚΕ για να ε, ξέρουμε και τη δική τους άποψη. Έχουμε τους επόμενους ομιλητές. Ντομινί Κρικέ είναι ο πρώτος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη, δημοσιονομικού, δημοσιονομικής φύσεως, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων για το πι γνωρίζουμε ότι θα λείπουν λίγο ε, γύρω στα 75 δις ε, υπό τις καλύτερες ε, προβλέψεις της Κομισιόν, αλλά μάλλον ακόμα χειρότερα τα πράγματα λόγω της αποχώρησης των Βρετανών φίλων. Άρα γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορεί να υπάρχουν νοπά χρήματα, φρέσκο χρήμα σε αυτό τον ε, μειούμενο προϋπολογισμό. Όμως, παρόλα αυτά, έχω και ένα ερώτημα να θέσω. Τι θα γίνει με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, διότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιέργως σε αυτές τις προτάσεις ε, ε μοιάζει και με βάση αυτά που μας είπε το Ινστιτούτο Μπρούγκελ, δηλαδή να στραφούμε κατά το εργατικό, στο, στο εργατικό δυναμικό και στην ε, μετατροπή ε, για να δούμε τι θα γίνει με επαγγέλματα που θα χαθούν και τι νέες δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν. Δεν μπορεί να αποκλειστεί τελικά εν μέρη να έχουμε έναν υποκανονισμό εφαρμογής ε, για να χρησιμοποιηθεί εν μέρη το ταμείο αυτό ε, και ίσως το ταμείο, το ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να χαθεί, άρα να χαθούν και κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής και να χαθεί και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό σας ευχαριστώ την προσοχή στα δημοσιονομικά θέματα και ακούγοντας τις ε, διάφορες παρεμβάσεις σκεφτόμουν ότι υπάρχουν κάποιες περιφέρειες της Ένωσης που ήδη έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κλεισίματος ε, ανθρακοριχείων στη Βαλονία, στο Βόρειο Καλέ, Πάντε Καλέ, κλείσανε ε, ανθρακοριχεία που ήταν η βάση της οικονομικής δραστηριότητας για τις περιοχές αυτές και όχι απλά κλείσανε αλλά πέραν όλων των άλλων κλάδων ε, έντασης ε, έπρεπε να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Πρώτον, το λουκέτο ε, στη, στα ανθρακοριχεία, δεύτερον, χαλιβουργία που έκλεισε και τρίτον, συναφή κλάδη που επλήγησαν. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει αλλού. Μπορεί να ήταν άλλες οι που επλήγησαν και άλλες οι εποχές τότε, όμως πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και ήταν πολύ σημαντικέ οι επιπτώσεις στην απασχόληση. Νομίζω ότι στις προκαταρκτικέ μελέτες ε, η Κομισιόν δεν κάνει καμία συσχέτιση με παρελθούσες ε, σχετικέ εμπειρίε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ω συντάξει γνωμοδότη από την Επιτροπή Τραν έχω να κάνω μια παρατήρηση. Στόχος αυτού του Ταμείου μετάβαση είναι το κλείσιμο θρακοριχείων ε, ή τέλο πάντων εκμεταλλεύσεων εξόριξη ορυκτών καυσίμων. Το καταλαβαίνω δεδομένη τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Δεύτερον, άλλο στόχο. Μετατροπή των βιομηχανιών ε, ή των κλάδων ένταση ε, άνθρακα ή ενέργεια. Παρόμοια αυτά τα δύο. Γιατί εκεί υπήρχαν πριν ε, ανθρακοριχεία και υπήρχαν και άλλε εξωτερικέ δραστηριότητε. Θέλω να επιστώ την προσοχή τη Επιτροπή Ρέτζη στο εξή το πρώτο αίτιο εκπομπών εξαιτία άνθρακα, που είναι και σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι μεταφορέ με 28% των εκπομπών. Και μετά έπονται βιομηχανία και στέγαση και θέρμαση. Και το 82% ε, προκύπτει από τη χρήση των κινητήρων, από τις οδικές μεταφορές και ιδίως σε περιοχές, περιφέρειες που θα θίγονται και από τα προβλήματα με το κλείσμα ανθρακοριχιών. 12 εκατομμύρια εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία των παροθερμικών κινητήρων που θα πρέπει να εκλείψουν με βάση τις προτάσεις σε 15-20 χρόνια ή τέλος πάντων θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή των συγκεκριμένων κινητήρων τα επόμενα χρόνια. Και επειδή υπάρχει ε, και η μεταφορά ε, προς την ηλεκτροκίνηση, 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν, θα θυσιαστούν. Φανταστείτε τι θα γίνει λοιπόν. Έχουμε και τις εξορρυκτικές βιομηχανίες, έχουμε τις βιομηχανίες έντασης άνθρακα. Όλα αυτά ε, σίγουρα σχετίζονται άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση. Γιατί αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τις εκπομπές διοξιδίου στις ε, στάθρα κορυχεία, εξωτικές ε, βιομηχανίες, ε, μεταφορές ε, ή, άλλοι κλάδοι, σε άλλους κλάδους έντας και ενέργειες, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και παντού προς Δυσμάς και προς Ανατολάς οι κλάδοι ε, της παραγωγής ε, θερμικών κινητήρων αντικατέστησαν ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις τις εξωτερικές δραστηριότητες. Άρα έρχεται τρίτη καταστροφή για αυτές τις περιφέρειες. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά, τις καταστροφικές δυνητικά επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά στην απασχόληση και στον κοινωνικό ιστό. Πρέπει να εστιάσουμε στους ανθρώπους, ε, στους εργαζομένους. Αλλά ε, νομίζω θα μείνουμε στα λόγια, γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα επίσης πρώτο επίπεδο εξόρυξη άθρακα, ένταση ενέργεια και θερμική κινητήρες. Αυτά τα τρία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, γιατί και το τρίτο, η σταδιακή κατάρριξη αυτών των κινητήρων θα έχει πραγματικά καταστροφικές επιπτώσεις. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρουσα παρέμβασή σου, Ντομινίκ. Εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών, πράγματι πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε στη, στον προβληματισμό μας όλες αυτές τις πτυχές. Ιδίω από τη στιγμή που θα γίνουν ταυτόχρονα όλες αυτές οι αλλαγές. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου αυτό νομίζω. Και παρακαλώ τον εισηγητή μας να συνεργαστεί στενά με τις ε, άλλες επιτροπές που θα ε, συνδεθούν σε αυτή τη διαδικασία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφο Ροβένα Πλούμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ερευνητικό Ίδρυμα, ε, από όλους τους προλαλήσαντες για τις συστάσεις τους, για όλους τους ομιλητές. Εκφράζω τη χαρά μου διότι η συγητή στην Επιτροπή των Περιφερειών είναι παρόν εδώ για το ίδιο ζήτημα. Έχουμε συναντηθεί, κύριε Δήμαρχε, και έχουμε ανταλλάξει τα νέα για το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Οφείλω να σας πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων για τον προϋπολογισμό. Πράγματι, τα χρήματα δεν φτάνουν. Μιλούμε για τα χρήματα τα οποία έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία μετάβασης, είναι, η οποία πρέπει να είναι δίκαιη, υπάρχουν. Ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ότι μπορεί να ενισχυθεί η εργασιακή διάσταση, η κοινωνική διάσταση. Μιλούμε για την προσέλκυση επενδύσεων. Και μιλούμε για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, ξέρετε, είναι ο βασικός πόρος και στη χώρα και στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις συστάσεις για το εργασιακό θέμα και για την σωστή κατανομή των κονδυλίων προκειμένου να υπάρξει επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ταμεία είναι παιχνιχρά. Το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά. Μου αρέσει η ιδέα της διάστασης του φίλου των δύο φίλων στο Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Μιλούμε για τις δεξιότητες, για τα προσόντα, για την απόκτηση νέων προσόντων και δεξιοτήτων ή για την ενίσχυση και αναβάθμιση των, ε, ε, των δεξιοτήτων. Μιλώντας για το κλάδο των μεταφορών, ξέρουμε ας πούμε ότι στους σιδηροδρόμους απουσιάζουν οι γυναίκες, δεν δουλεύουν αρκετές γυναίκες και ότι πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών εργαζομένων σε αυτό το κλάδο. Σε αυτές τις ανθρακοπαραγωγικές περιοχές που είναι σε μετάβαση το ίδιο ισχύει. Άρα και με την εποχή της ψηφιοποίησης μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Η εποχή της ψηφιοποίησης παρέχει ευκαιρίες να εμπλέξουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτό το εγχείρημα και χαιρετίζω αυτή την ιδέα για τη διάσταση των φύλων. Και όταν γίνεται λόγος για ε, την κοινωνική εργασιακή αυτή διάσταση, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία που έχει η επιλεξιμότητα ή μη ορισμένων project. Για παράδειγμα, αποκλείονται όλες οι επενδύσεις που ε, σχετίζονται με τις κοινωνικές υποδομές και όχι μόνο. Θέλω όμως να σας μιλήσω για αυτές τις κοινωνικές υποδομές. Δηλαδή, οι επενδύσει που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να υπάρχουν οι ακατάλληλες υποδομές. Εάν τώρα οι κατάλληλες υποδομές δεν παρέχονται βάσει του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι χρειάζεται ξεχωριστή προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα και ο διαχωρισμός των ενσωματωμένων και μέτρων θα εμφανίζεται στο Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση όπως αναφέρεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τα διαβάζω αυτά για την παρακολούθηση της συζητήσης. Θέλω λοιπόν να πω στο δόκτωρα ε, κύριο Τζίμα από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, το Joint Research Center, ότι η πλατφόρμα για τις ανθρακοπαραγωγικές περιοχές που είναι σε μετάβαση την οποία πλατφόρμα ξεκίνησε μαζί με εσά ο Επίτροπος Μαρουσεύσκεβιτς πρόπερση, ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία, με πολύ καλά αποτελέσματα, για τη Ρουμανία για παράδειγμα, γιατί τώρα προετοιμάζουμε αυτή τη στρατηγική για μία από τις βασικές ανθρακοπαραγωγικές περιοχές που θα υποστεί αυτή τη μετάβαση και θα διέλθει από αυτή τη μετάβαση. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε για να υπάρξει μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Θα υποβάλουμε τις τροπολογίες έγκαιρα και θα διαβολευτούμε με τους συναδέλφους, με τον συνάδελφο από την Επιτροπή των Περιφερειών και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, cher collègue. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Αμαρού έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω στα πορτογαλικά, τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ θερμά, με κάθε ειλικρίνεια, για τη διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου, για την ε, φιλοξενία αυτής της συζήτησης, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους σκιώδεις εισηγητές και ε, την προσοχή του εισηγητή στο γεγονός ότι όλοι εσείς έχετε δουλέψει εντατικά και παραμένει ε, εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί και ο ρυθμός πρέπει να παραμείνει εντατικός. Ξέρετε, εγώ όταν εξελέγει, όταν ήρθα εδώ, ήταν ένα θέμα που με απασχολούσε πολύ. Ήρθα λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση λίγο καθυστερημένο και δεν γνωρίζω εάν κατάλαβα πολύ καλά, εάν κάτι έχασα. Πρόκειται για δράσεις, για πρωτοβουλίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσε, φιλόδοξε, που έχουν ως στόχο ε, κάτι το οποίο είναι πολύ ενάρετο και ε, το, στο οποίο προσυπογράφουν όλοι και από την αριστερά και από τη δεξιά. Να έχουμε μια Ευρώπη δυνατή δηλαδή και αλληλέγγυα. Όμως, εμείς που επίσης συμμετέχουμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαμε εκεί εδώ, γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Μιλούμε για το πρόγραμμα από την εκμετάλλευση, την αγροτική μέχρι και το πιάτο. Ε, μία ενιαία δηλαδή προσέγγιση. Είναι αξιοπρόσεκτο το πρόγραμμα αυτό. Ε, έχω όμως να πω ότι αν τελικά δεν θέλουμε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη, ε, τελικά δεν θα κατασκευαστούν ούτε πυρούνια και ούτε πιάτα για να φάει κανείς, γιατί θα λιμοκτονήσουμε και δεν θα έχουμε τίποτα να φάμε ούτως ή άλλως. Όλοι συμφωνούμε με αυτή τη νέα πράσινη συμφωνία. Και τι κάνουμε όμως παρόλα αυτά, κάνουμε περικοπές στη γεωργία. Επειδή συμφωνούμε με αυτή τη φιλοδοξία και αυτό το στόχο, τον καθόλου ενάρετο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σκεφτόμαστε τον τοπικό πληθυσμό. Δεν θα σκεφτόμαστε τις περιφέρειες. Δεν θα ε, σκεφτόμαστε την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριε Πρόεδρε, ένας μέγας ειδικό είπε κάποια στιγμή ότι οι περιφέρειες που θέλουν να πάνε προς την ε, απανθρακοποίηση, αν θέλετε, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ε, θα πρέπει να υποφεληθούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Αλλά μπορεί να μην υπάρξει καν Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γιατί μπορεί να είναι επιλέξιμες οι δράσεις για την απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, αλλά με άλλο τρόπο επιλέξιμες. Ε, πρέπει όλα αυτά να τα κατασυγάσουμε, εάν θέλουμε μόνο να κάνουμε μάρκετινγκ να επινοήσουμε ένα πρόγραμμα πολύ ποιοτικό και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει τι ωραία που είναι αυτά, ας ε, ε, συνάψουμε αυτή την ε, ευτυχή συμμαχία, αλλά πληρώστε εσείς γιατί εμάς τα ταμεία μας είναι άδεια. Ξέρετε, στα πορτογαλικά έχουμε μια έκφραση, λέει ο λαός, ότι είναι λίγο σαν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Μας δίνεται από το ένα χέρι αυτό που μας παίρνετε από το άλλο χέρι να ένα τέλειο πρόγραμμα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εποχές, ε, εκπομπές, αλλά ειδού λιγότερα χρήματα για την κοινή αγροτική πολιτική και λιγότερα χρήματα για την συνοχή. Πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Εγώ νιώθω χαμένο μέσα σε αυτόν τον ωκεανό. Όλα αυτά στερούνται νοήματος. Είναι άνευ νοήματος και το λέω με, με όλο το σεβασμό που τρέφω προ το πρόσωπό σας. Υπάρχει άρρηκτος δεσμός με την οικονομία. Ε, δεν πρέπει να έχουμε αποκλεισμό ούτε εγκατάλειψη. Έχουμε μια εργασιακή και κοινωνική τόσα, η οποία πρέπει να είναι παρούσα μαζί με ένα πολύ ισχυρό στοιχείο ανάπτυξης. Και αυτό πρέπει να είναι παρόν. Και κάτι που μου διέφυγε να σας πω είναι και το εξή. Δεν είμαι ευρωβουλευτής εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά ε, και στην Πορτογαλία και αλλού ε, και στις άλλες χώρες λέμε ότι το θέμα είναι η πολιτική. Για πολιτική μιλάμε. Εάν λοιπόν ε, υψώσουμε το πύχη, αν έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες, και εγώ τις έχω και τις τρέφω, δεν θέλω να απογοητευτώ τελικά στο τέλος και δεν πρέπει κανείς μας να απογοητευτεί. Και γι' αυτό και απευθύνω αυτή την έκκληση. Μία Ευρώπη φιλόδοξη και μία Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλόδοξη, η οποία θα θέτει ξεκάθαρους στόχους. Ε, τι κάνει τελικά, τα λέει αυτά στα λόγια και τελικά πνίγει το πρόγραμμά της με την ελληπή χρηματοδότηση που δέχεται. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά αμφίσιμα δεν πρέπει να υιοθετήσουμε τη γλώσσα της αμφισημίας, αμφισημίας, να αγωνιστούμε για μια πιο πράσινη Ευρώπη, πιο υγιή Ευρώπη, αλλά με ισχυρή παραγωγή και ισχυρή εργασιακή συνιστόσα. Και γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο παρουσιάζει ελλείψεις σημαντικές και υστερεί ε, σε σχέση με τις φιλοδοξίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Καρβάλάης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να μιλήσω πορτογαλικά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τους προλαλήσαντες στο σύνολό τους για την πολύ σημαντική συνεισφορά τους στη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την εξής ανησυχία που έχουμε. Από ό,τι φαίνεται επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια επιχειρήματα. Παρόλα αυτά, εάν δεν καταλαγιαστούν οι ανησυχίες μας, το μόνο που θα κάνουμε είναι να ευθύνουμε συνεχώς τα ίδια ερωτήματα τα οποία παραμένουν κρίσιμα και επίκαιρα ε, περισσότερο σήμερα παρά ποτέ. Η υποχρέωση ηθική και δοντολογική είναι η μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλό ενεργειακό αποτέλεσμα αποτύπωμα, με ουδέτερο ενεργειακό και κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι υποχρέωσή μας αυτή έναντι του πλανήτη στον οποίο διαβιούμε. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια μετάβαση δίκαιη, ισορροπημένη, η οποία να μην θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία της πράσινης συμφωνίας, η οποία να μην οδηγεί σε κατακαιρματισμού, σε ρογμή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και γι' αυτό όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές η μετάβαση αυτή πρέπει να πλησιώνται, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και εργαλεία. Να με διορθώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν σφάλω, όμως από ό,τι φαίνεται αυτό που έχουμε επιτάπητος είναι πρόθεση των κρατών μελών να μετατρέψουν τη χρηματοδότηση του Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση σε χρηματοδότηση που θα προέρχεται από το Ταμείο για τη Συνοχή. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Αλλά φαίνεται ότι μειώνουν τις πιστώσεις για την πολιτική συνοχής και τα κράτη-μέλη όπως η Πορτογαλία, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, δεν το λέω για να υπερασπιστώ τα εθνικά μας δίκαια αν θέλετε, καθόλου. Ε, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες δεν βασίζουν την οικονομία τους σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα και στην παραγωγή αυτού. Και γι' αυτό έχουν πολύ μικρότερη παρουσία στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Όμως υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια μεταστροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τη γνώμη μου, στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο οι χώρε αυτέ θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερε δυσκολίε. Σω δεν γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση, γιατί είναι η πρώτη κοινοβουλευτική μου θητεία, ούτε έξι μήνες δεν είμαι εδώ, ίσως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά, αλλά το θεωρώ άδικο. Είναι μια διαδικασία άδικη αυτή, η υπόθεση χώρε να έχουν ε, επενδύσει και να μεταστραφεί στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τελικά να χάσουν χρήματα από το Ταμείο συνοχή και να μην τα πάρουν το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση γιατί δεν εξαρτώνται ιδιαίτερα από τον άνθρακα. Νομίζω ότι δεν καλλιεργείται έτσι η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και αυτό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Το έχουμε δει την τελευταία δεκαετία και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει πλήγμα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και το ευρωπαϊκό όραμα γενικότερα. Ευχαριστώ. Αυτό ακριβώ είναι ο στόχο τη συνεδρίασής μα, να τεθούν οι ερωτήσει. Όταν δεν έχει κάποιο καταλάβει καλά ή λοιπόν πληροφορίε, γι' αυτό πρέπει να γίνει η δύσκολη αυτή δουλειά σίγουρα, αλλά παρακαλώ να σημειώνετε τις ερωτήσεις. Ε, στρέφομαι προς την Κομισιόν για να μπορέσετε να μας απαντήσετε στο τέλος. Ο πρώτος αντιπρόεδρος μας τώρα έχει το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι ακριβής, γι' αυτό θα μιλήσω πολωνικά. Το Green Deal είναι ένα γεγονός, είναι κάτι το πραγματικό. Δεν θα πρέπει να το συζητάμε πια. Πιστεύω επίσης ότι χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους, μεγαλειώδεις στόχους θα έλεγα. Και αυτή η συμφωνία, αυτό το σχέδιο μάλλον, που αναφέρεται ως Green Deal ε, στις ημέρες μας είναι πραγματικά ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δυστυχώς άκουσα κάποια σχόλια που με κάνουν ε, να ανησυχώ για το πώς πρόκειται να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και ποιο θα είναι το τίμημα. Γιατί από ό,τι μόλις άκουσα, καταρχάς άκουσα κάτι που το ξέρω εδώ και αρκετό καιρό, ότι δηλαδή η είναι η πολιτική συνοχής που σε μεγάλο βαθμό θα, χρηματοδοτη... θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς, στις επιχειρήσεις, ε, σε άλλους φορείς που δεν έχουν πολύ σχέση με τη μετάβαση. Και αυτό σημαίνει αποδυνάμωση, ε, διάλυση θα έλεγα στο μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής που έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με την κοινή αγροτική πολιτική. Έχω και έναν άλλο φόβο που πρέπει να σας ομολογήσω και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση που απλώς δεν αρκεί για να καλυφθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Ίσως ε, θα επαρκέσει μόνο για να καλυφθεί η κοινωνική διάσταση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πού θα βρεθούν τα χρήματα για τους άλλους τομείς που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα από την κοινωνική πολιτική, ε, από συνοχής. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρετηθουν ε, από άλλα πράγματα που θα έκαναν με τα χρήματα αυτά και δεν είμαι σίγουρος αν αυτή είναι η σωστή λύση. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση, να είμαστε όλοι πιο ρεαλιστές και πιο συγκεκριμένοι. Μιλάμε για το μέλλον μας και όχι για κάτι το αφηρημένο λέμε ότι τα θρακοριχεία θα μπορούσαν να γίνουν ε, τουριστικά αξιοθέατα και μουσεία. Μα πόσα μουσεία χρειαζόμαστε ε, σε τελευταία ανάλυση και ειδικά τέτοια μουσεία. Και μάλιστα τέτοια μουσεία ίσως υπάρχουν ήδη σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ε, στους ανθρώπους αυτούς που θα χάσουν τις δουλειές τους, τι να τους πούμε, ότι θα γίνουν ανεξάρτητοι επαγγελματίες, θα δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις Ταυτόχρονα έχουμε στοιχεία που ε, μας δείχνουν ότι 80% των ε, δημιουργούμενων επιχειρήσεων ε, κλείνουν, φαλυρίζουν μέσα στο πρώτο χρόνο της ύπαρξής τους. Πώς θα τα επιτύχουμε λοιπόν όλα αυτά που θέλουμε, πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε, γιατί προς το παρόν και λυπάμαι που το λέω, αλλά όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, δεν έχουμε ε, τίποτα άλλο να απαντήσουμε σε αυτό παρά μόνο το ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τον άνθρακα. Εντάξει, αλλά δεν προτείνουμε καμία εναλλακτική για αυτούς τους ανθρώπους που θα τους χτυπήσει σκληρά αυτή η μετάβαση. Όπως είπαν πολύ σωστά οι ομιλητές, εκατοντάδες, οι, που κάνανε τις παρουσιάσεις, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ε, θα πληγούν από αυτή τη μετάβαση. Δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να μεταφερθούν σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό, γιατί είναι άσχημο, γιατί δεν ξέρω εγώ τι και πρέπει να χτίσουμε ένα καινούριο σπίτι. Εντάξει, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πληρώσουμε είναι τα θεμέλια αυτού του σπιτιού και τίποτα παραπάνω. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Αντιπρόεδρε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές ε, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Ε, θα ήθελα Καταρχά να πω ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένο με καλές προθέσεις. Και στην κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με αυτή την πρόταση τη Κομισιόν, δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε, να την αφήσουμε σε εκκρεμότητα ή να την απορρίψουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι χρήματα θα είναι διαθέσιμα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουμε τα χρήματα για να χτίσουμε αυτό το σπίτι ε, που ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Αυτά τα 7,5 δις που ακούστηκαν σήμερα το απόγευμα και τα ακούμε εδώ και πολύ καιρό πια, υποτίθεται ότι θα έρθουν επιπλέον του προϋπολογισμού. Όμως τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμφωνήσει καν για το συνολικό χρηματοδοτικό ε, φάκελο. Ε, πού θα κοπούν αυτά τα χρήματα από τη συνοχή, από τη γεωργία που ήδη ε, το παλεύουν. Ε, ας είμαστε απολύτως ε, ξεκάθαροι στο σημείο αυτό. Και μιλάμε για την κοινωνική διάσταση. Μιλήσαμε πολύ για την κοινωνική διάσταση. Φυσικά και είναι πολύ σημαντική. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να εξασφαλίζουν το προστοζή. Αλλά στις διαφάνειες που είδαμε, σήμερα ε, γίνεται λόγος για περιοχές ε, ε, εξόριξης λοιπά με τα ορυχεία, αλλά δεν μιλάμε για συναφείς δραστηριότητες που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα ενός ορυχείου. Τι θα γίνει άμα κλείσει ένα ορυχείο. Στην Ρουμανία, παραδείγματο χάρη, 3,7% της ισχύω στο δίκτυο προέρχεται από την εξορυκτική βιομηχανία με τι θα αντικατασταθεί αυτό. τι χρειαζόμαστε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια. Από πού θα τη βρούμε, με τι, από πού θα την αντικαταστήσουμε όταν θα χαθεί. Δεν θα έχουμε συνεχώς ούτε ε, ε, αιωλική ε, ενέργεια, ούτε ηλιοφάνεια. Από πού θα τη βρούμε αυτή την ηλεκτρική ισχύ που θα λείψει. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται λόγος για το φυσικό αέριο, που μπαίνει, εντάσσεται και το φυσικό αέριο ε, στη συζήτηση για την μετάβαση. Θα συνεχίσουν να επενδύσει στο κλάδο αυτό ή θα σταματήσουν. Η πυρηνική ενέργεια. Θα συνεχιστούν αυτές οι εξελίξεις ή θα ε, σταματήσουν. Γιατί η βασική ερώτηση είναι από πού θα βρούμε την ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον. Πώς θα γίνεται η παραγωγή αυτής της ισχύω που χρειαζόμαστε στο μέλλον. Και θα επενδύσουμε στις τεχνολογίες που ε, σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πρώτα και μετά να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις εκπομπές. Δεν μπορούμε να παίζουμε το Θεό, δεν είμαστε θεοί. Ε, πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Ε, ποιος θα είναι ο επόμενος ε, κλάδος που θα ε, γίνει στόχος της Κομισιόν μετά τα ορυχεία και την εξορυκτική βιομηχανία. Τι θα γίνει με αυτούς τους άλλους τομείς. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να ε, σκεφτούμε το θέμα της χρηματοδότησης. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα και με ποιους εναλλακτικού τρόπους θα γίνει η παραγωγή της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χαθεί έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σολής Περέση. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους του εισηγητέ, τους εμπειρογνώμονε ε, που μας μίλησαν για το Ταμείο δίκαιη Μετάβασης και να πω ότι νομίζω ότι συμμερίζομαι με τους συντρόφου και τις συντρόφισες της ανησυχίας μας για το Ταμείο αυτό. Είναι αναγκαίο σίγουρα αν θέλουμε ευρωπαϊκές περιφέρειες να προχωρήσουν προς μια ενεργειακή μετάβαση και μια οικονομία χωρίς άνθρακα και σίγουρα χρειάζεται βοήθεια ε, στις περιφέρειες μέσω αυτού του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης που όμως το πρόβλημα ποιο είναι ότι δεν είναι δίκαιο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή τιμωρεί το Ταμείο τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που έκαναν ε, αυτό που πρέπει. Και θα σας δώσω το παράδειγμα της Ισπανίας. Η δική μου περιφέρεια, η Αστούρια, οι άλλες περιφέρειες ε, που είδαμε και στους χάρτες, στις παρουσιάσεις Αραγών, Καστήλη, Λεών, έχουν κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες κυρίως ε, παραγωγές, περιοχές, ιδίως η δική μου. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κλείσουν ανθρακορυχεία. Πέρυσι έκλεισε και το τελευταίο ανθρακορυχείο και σήμερα έκλεισαν, γιατί ε, να κλείνουν και οι μονάδες παραγωγής ε, θερμοελεκτρικής ενέργειας. Κλείνουνε. Όλα αυτά επηρεάζουν όμως σημαντικά την ανεργία που αυξάνεται και κυρίως μεταξύ των νέων. Και το αποτέλεσμα είναι και απερίμωση των περιφερειών αυτών. Επομένως, Πολύ θα χαιρόμουν να πιστέψω ότι πράγματι θα πάμε σε αυτή τη δίκαιη μετάβαση που δεν θα επηρεάσει αρνητικά τον πληθυσμό για την απασχόληση, όμως το έχουμε δει ξεκάθαρα στη χώρα μου τι αποτέλεσμα είχε. Γι' αυτό ζητώ το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης να λάβει υπόψη κριτήρια απερίμωσης, κριτήρια ανεργίας και ανεργία των νέων μεταξύ άλλων, και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περιφέρειες που έκαναν αυτό που έπρεπε και παρόλα αυτά τιμωρούνται. Κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η φιλοδοξία. Δηλαδή, αυτά τα ταμεία και τα κοντήλια πρέπει να συνδέονται με σαφείς δεσμεύσεις ε, προς ε, κλιματική μετάβαση και απαλλαγής από τον άνθρακα. Επίσης, λέμε ότι τα μειοδικές μετάβασης ε, και τα, το, ΕΤΕΠ, το ΕΤΠΑ, υπάρχει αλληλεπικάλυψη πολλές φορές μεταξύ αυτών των δύο ταμείων. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα κονδύλια του, του ΕΤΠΑ. Ε, όλοι ανησυχούμε που βλέπουμε μειώσεις, περικοπές στην πολιτική συνοχή. Και σίγουρα το Ταμείο Δίκαιος Μετάβαση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την απώλεια. Και συμμερίζομαι τις ανησυχίες όλων όσοι έλαβαν πριν από μένα τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κρυκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος του Ταμείου είναι να ε, διευκολύνει τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής μετάβασης. Ο πρόεδρος πολύ σωστά το έθεσε. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε, πόσο θα επιτύχουμε στο στόχο αυτό. Θα μπορέσουμε όμως να επιτύχουμε το στόχο αυτό μόνο με 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχετε, έχει τεθεί πολλές φορές αυτό το ερώτημα και θεωρώ, όπως και πολλοί άλλοι, ότι είναι πολύ μικρό αυτό το ποσό, πολύ ταπεινό. Και με τέτοια ποσά δεν μπορούμε να ε, έχουμε ένα πραγματικό αντίκτυπο ε, στο θέμα της μετάβασης. Ε, υπάρχει βέβαια και το θέμα των δανείων, της ε, εθνικής συνεισφοράς, της ε, συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα και ε, επίσης γίνεται λόγος για μεταφορά από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ μια μισή ως τρεις φορές του ποσού του Ταμείου Μετάβασης. Όμως οι πόροι που θα έχουμε στη διάθεσή μας ήδη θα είναι μειωμένοι σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αν μειωθούν περαιτέρω, θα είναι πολύ δύσκολο για τις περιφέρειες και για τα κράτη να ε, εκπληρώσουν τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Επίσης, η τεχνολογική ουδετερότητα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ιδιαίτερα, αν λάβουμε υπόψη μας ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2019. Τα κράτη-μέλη πρέπει να σκεφτούν ε, τι θα κάνουν σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλη συνεξάρτηση ε, όπως είναι η Πολωνία μαζί με, όπου υπάρχει εξάρτηση και από το φυσικό αέριο και από την πυρηνική ενέργεια. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της μετάβασης. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σαφές από αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω η Κομισιόν να είναι ανοιχτή για αλλαγές, γιατί πραγματικά πολλές αλλαγές θα χρειαστεί να επέλθουν για να είναι αποτελεσματικό αυτό το νέο ταμείο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. στα πλαίσια του ανηλαιού ανταγωνισμού των κολοσσών της ενέργειας και των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, δίκαιη μετάβαση για τους λαούς δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει. Αν θέλετε αυτό το δείχνει και η εμπειρία συνολικά και πολλών λαών της Ευρώπης αλλά και του λαού της Ελλάδας, της χώρας μου. Ιδιαίτερα η εμπειρία που έχουν οι κάτοικοι των περιοχών που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν συνδεθεί με την παραγωγή ηλεκτρενέργειας στη χώρα και στη Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία και αλλού. Γιατί, γιατί η πολιτική την οποία σήμερα έχουμε φτάσει να, μας, να ονομάσουμε δίκαιη μετάβαση Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal δεν εμφανίστηκε από μόνη της. Έρχεται σαν συνέχεια. Έρχεται σαν συνέχεια, για παράδειγμα, τη πολιτική απελευθέρωση του κλάδου τη ενέργεια, που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 90, το 2000, την εφάρμοσαν όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει, όπου ξεπουλήθηκε σιγά σιγά η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού υπήρχε. Μπήκαν οι ιδιώτε, μεγάλα μονοπόλια στο παιχνίδι. Ποιο πλήρωσε το μάρμαρο, ο ελληνικός λαός με αυξήσει στα τιμολόγια. Στη συνέχεια, με τις ευνοϊκές ρυθμίσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σπρώξει μεγάλες, ε, μεγάλους τεχνολογικούς ε, ε στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών, Ποιο πλήρωσε πάλι το μάρμαρο, φορτώθηκε ο ελληνικό λαό με πράσινου φόρου, με ενισχύσει για τι ΑΠΕ, εκατοντάδες ευρώ, για να μην πω χιλιάδε στον ετήσιο προπολογισμό του. Και σήμερα, με τη λογική της απολιγνητοποίηση, αντίθετα με τη λογική του πώς δίκαια να μεταβούμε, τι έχουμε, έχουμε κλείσιμο βασικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από λιγνίτη. Δεν λέμε εμείς ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος, όμως μπορεί σήμερα ένα διαφορετικό μείγμα, το οποίο θα το ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιοποιήσεις το προϊόν που έχεις από τη χώρα σου με νέους, νέες μονάδες συνδυασμένου κύκλου με χαμηλούς ρήπους περιβαλλοντικά έτσι ώστε να μπορέσεις σε ένα διάστημα να ρυθμίσεις καλύτερα το μείγμα. Γι' αυτό και αντιδρά συνολικά ο λαός των περιοχών εκείνων είναι σήμερα σε κινητοποίηση, ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που εφάρμοσε πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιδρά και απορρίπτει αυτά τα σχέδια. Το θέμα είναι υπάρχει λύση, υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Γιατί υπάρχει και η τεχνολογία σήμερα, υπάρχει και η επιστημονική γνώση να τα συνδυάσει. Αυτό που δεν υπάρχει όμω, κατά την άποψή μα, είναι δεν υπάρχει ένα ενιαίο κρατικό φορέα ενέργεια, ο οποίο να μπορέσει αξιοποιώντα του πόρου που έχει στο έδαφο του να σχεδιάσει την παραγωγή ηλεκτρενέργεια, να μην ενταθεί η ενεργειακή εξάρτηση, για παράδειγμα, από το φυσικό αέριο, το οποίο θα αναγκάζεσαι να το αγοράζει από τρίτε χώρε, δεύτερε χώρε, το οποίο σου δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να παρέχει φτηνό ρεύμα για τι λαϊκέ οικογένειε και ταυτόχρονα να καλύπτεις την ανάγκη τη βιομηχανική παραγωγή τη χώρα στην πορεία αλλαγή του μείγματο, έτσι ώστε να γίνεται συνεχώ καλύτερο και φιλικότερο προ το περιβάλλον. Βεβαίω, για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα διαφορετικού τύπου σχεδιασμό και μέσα στο εσωτερικό τη χώρα, ένα επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό τη οικονομία, όπου σε αυτά τα πλαίσια μπορεί πραγματικά να λύσει και το ζήτημα τη ενέργεια συνολικά σαν λαϊκό αγαθό χωρίς να φορτώνει συνέχεια και κακής ποιότητας υπηρεσίες και ενεργειακή φτώχεια το λαό και βεβαίως να μην κρέμεται και πάνω από το κεφάλι του σαν δαμόκλεια σπάθη όπως λέμε στην Ελλάδα η απειλή να του πάρουν το σπίτι στους πληστηριασμούς ακόμη και για το ποσό των 500.000 ευρώ ε, χρέη προς την εταιρεία ηλεκτρισμού ενώ ταυτόχρονα να αφήνονται ασίδωτα να δρουν και να χρωστούν οι μεγάλοι οφειλέτες, οι μεγάλες εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστούμε. Α. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφος Πεκάρη να ανοιχτεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω φιλανδικά, αν το προσέξατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να πω δύο λόγια όμως. Και αυτό γιατί θέλω να σας επισημάνω ότι η τύρφη είναι από εντελώς. Εμείς είχαμε 100.000 εκτάρια τύρφη στη Φιλανδία. 20 τεραβάτ ενέργειας παράγουμε με τη χρήση της τύρφης κάθε χρόνο. Δηλαδή δύο φορές ε, την ενέργεια που χρησιμοποιεί όλο το χρόνο η Ιστονία. Η τύρφη είναι ορυκτό καύσιμο. Και θα πρέπει και αυτή σιγά σιγά να εγκαταλειφθεί. Ε, εγώ θέλω να ληφθεί υπόψη η τύρφη στην έκθεση. Μιλάμε για τεράστιες ε, περιοχές, τρυφώδεις περιοχές στη χώρα μας. Αυτό ήταν το σχόλιο και έρχομαι στην ερώτηση που ήθελα να διατυπώσω. Έχουμε τους κανόνες περί ενισχύσεων. Στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης υποτίθεται πρέπει να τηρούνται πολύ αυστηρά. Τι θα πει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα περιφερειακά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και υπάρχουν κάποια όρια στι ποσοστιαίες μονάδες, Παραδείγματο χάρη στη Φινλανδία. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη. Αλλά δεν μπορεί να δοθεί ενίσχυση ε, λόγω των κανόνων περί εθνικών ενισχύσεων. Τι γίνεται με τις δημόσιες συμβάσεις, τις δημόσιες προμήθειες ε, που θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν για την ε, αναζωογόνηση των περιοχών που πλήττονται. Λαμβάνετε αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, πολλά τα ερωτήματα θα πρέπει και αυτό που είπατε να μας απασχολήσει. Όταν ε, θα έρθει η στιγμή της εξέτασης της έκθεσης του συναδέλφων Στέφαν Μπιζού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους για τις πολύ ποιοτικέ παρεμβάσεις. Άκουσα πολλές ανησυχίες να εκφράζονται. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο της ανταλλαγής απόψεων να ανοίξουμε την πόρτα στην αισιοδοξία. Ναι, είναι πολύπλοκο σίγουρα να εξευρεθούν λύσεις για να είναι επιτυχημένη η ενεργειακή αυτή μετάβαση. Και γνωρίζουμε ποιε είναι οι προκλήσεις, τι διακυβεύεται, ποιε είναι οι δυσκολίες. Το είδαμε και ακούσαμε στις παρεμβάσεις τίθεται το θέμα των ΑΠΕ. Προς ε, Δυσμάς Ανατολάς, ε, Βορρά και Νότο αναζητούνται εναλλακτικέ για τη, αντί της χρήσης του άνθρακα. Παίζουμε το χαρτί της αιωλικής, της ηλιακής ενέργειας. Αναζητούμε λύσεις για την Ευρώπη του αύριο. Και πρέπει να σας πω όμως ότι ήδη υπάρχει και στην Ευρώπη του σήμερα ε, αυτή η εναλλακτική λύση. στις, στα γαλλικά υπερπόντια δάφη και διαμερίσματα. Γίνονται πάρα πολλά. Επίση, στα Κανάρια νησιά ε, έχουμε ενεργειακή αυτονομία σε μεγάλο βαθμό ε, με τα αιωλικά πάρκα. Στι Αζόρε, επίση, για θερμική ενέργεια. Πρέπει να έρθετε λοιπόν στα υπερπόντια δάφη και διαμερίσματα Γαλλία και άλλων χωρών για να δείτε τι εναλλακτικέ υπάρχουν στο πλαίσιο των ΑΠΕ. Με έχετε ακούσει συχνά να το λέω η Ευρώπη είναι μια ευκαιρία για τα υπερπόντια εδάφη. Αλλά να που για την περίπτωση της αναζήτησης εναλλακτικών, τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη είναι η λύση για την Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ροπέ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, Θέλω η Κομισιόν να προσέξει την εξή πτυχή. Μας υποβάλλατε εδώ μια έκθεση. Τη Λιθουανία όμως τη βάζετε στις περιοχές ΝΑΤΣ 2. Αυτό έγινε το 2016. Και νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Γιατί είναι ένα σοβαρό σφάλμα που πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον σε ό,τι αφορά το Ταμείο Δικής Μετάβασης. Έχει δοθεί τον αρκτήριο λάκτισμα και πρέπει αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε να είναι ευεργετική για την Ένωση συνολικά. Το ίδιο ισχύει όμως και τις αμονωμένες περιφέρειες. Η Κομισιόν έχει θέσει φιλόδοξους στόχους, όμως τι γίνεται με τον προϋπολογισμό. είναι, κινείται ακόμα στη σφαίρα της φαντασίας ο προπολογισμό. Δεν έχουμε ακόμη ένα πι και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιε είναι οι χρηματοδοτικέ δυνατότητε και μακροπρόθεσμα. Δεν μιλάω μόνο για την επόμενη επταετία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε σοβαρέ επενδύσει. Τι έχει να πει από αυτό η Κομισιόν. Επίση, πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στην υφιστάμενη εμπειρία. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μπήκε λουκέτο σε πυρηνικά εργοστάσια. Οι τοπικές αρχές έπρεπε να αντιμετωπίσουν ε, τεράστια προβλήματα και τα αντιμετώπισαν με επιτυχία. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτές τις εμπειρίες να τις ε, λάβουμε υπόψη. Στη Λουθάνία έχουμε παρόμοια εμπειρία, διότι παροπλίζουμε και εμείς ε, το πυρηνικό μας εργοστάσιο θα ήθελα να τονίσω ότι σε τέτοιες ε, περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες, γιατί μόνο αν έχει γίνει καλή προετοιμασία εκ των προτέρων, τα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να είναι μικρότερα. Εξετάζεται το πρόβλημα και οι πόλεις της Οπότε κανείς βλέπει τι ε, προβλήματα θα προκύψουν, παραδείγματο χάρη, για την επόμενη 15 ετία. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα. Υπάρχουν ίσως ε, κάποια προγράμματα εισαγών-εξαγωγών που μπορούν να προωθηθούν ε, η, η παραγωγική δυνατότητα, ικανότητα να προσανατολιστεί σε κάποια συγκεκριμένα αγαθά κτλ. Οπότε δεν θα είναι η μόνη εναλλακτική για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιφέρειες να εγκαταλείψουν την περιοχή που ζουν και να πάνε αλλού, να αναστήσουν την τύχη τους. Άκουσα πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες από τους συναδέλφους, αλλά για να γίνουν όλες πραγματικότητα πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να κλείσω τον κατάλογο. Ζαλεύσκα και Τζόρτζιαν αν με καλά, είναι οι επόμενοι ομιλητές. Komisji Środowiska i tam takiej refleksji gospodarczej absolutnie nie ma. Powtarzane są tutaj zdania, że Zielony Ład jest faktem. Nie, on nie jest faktem. On na razie jest celem. Υπάρχει ένας στόχος. Υπάρχουν ιδέε, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι σαν να παίρνουμε ένα τρένο, αλλά δεν ξέρουμε πού είναι ο σταθμός και δεν έχει και γραμμές να τρέξει το τρένο. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε πάνω σε τέτοιο τρένο. Ξέρουμε μόνο που θέλουμε να πάμε, τίποτα άλλο. Λείπει μία πλαισίωση γενικότερη αυτής της πρότασης. Ε, πρέπει να δούμε τη γεωργία, την ενέργεια, τις εκπομπές. Όλα αυτά δεν υπάρχουν μέσα στον κανονισμό. Δεν κοιτάμε την οικονομία γενικότερα στο σύνολό τη, κοιτάμε μόνο το Green Deal. Στην Πολωνία, στο παρελθόν, έχουν κλείσει ορυχεία. Στην περιοχή εκείνη όπου έκλεισαν τα ορυχεία. Έχουμε ε, μια οικονομική κατάσταση κάτω του μέσου όρου φυσικά. Ε, έχουν επενδύσει, ήδη η πολωνική κυβέρνηση ε, επένδυσε στην περιοχή αυτή. Εδώ τώρα μιλάμε για 7,5 δισεκατομμύρια και θεωρούμε ότι αυτό είναι ε, ένα κίνητρο αρκετό για να προσελκύσουμε και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια. Είναι αυταπάτη αυτό το πράγμα. Ρωτήστε τα κράτη-μέλη, εμείς θα σας πούμε πόσα χρειαζόμαστε. Όλα αυτά πρέπει να υπολογιστούν ε, από τους υπουργούς Μόνο ακούγοντάς τους ε, οι, οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών, μόνο αυτοί μπορούν να κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια παράλογη κατάσταση. Μιλάμε για κατάργηση κάποιων μέσων μεταφοράς και αύξηση των εκπομπών σε 3 εκατομμύρια τόνους διεξουδίου του άνθρακα, ε, δημιουργία νέων θέσεων ε, στάθμευσης, ε, κόψιμο των δέντρων, δηλαδή η Κομισιόν δεν μιλάει με εμάς, μιλάει και κλείνει συμφωνίες με την Μερκοσούρ λέμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές των ενεργοβόρων κλάδων της βιομηχανίας και τι κάνουνε ε, αυτές μεταφέρονται στην Κίνα παραδείγματος χάρη Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο αλλά ε, Πραγματικά ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους για την πολύ ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ εσείς, αγαπητέ συνάδελφοι. Όχι, όχι, από πίσω. Ο από πίσω σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω τις αμφιβολίες μου σε σχέση με το πεδίο αυτού του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Δεν υπάρχουν καν απαιτήσει για την τεχνολογική ουδετερότητα. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες αποκλείονται, αλλά τις οποίες χρειαζόμαστε αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση. Και δεν είναι δικαιολογημένη η έλλειψη αυτών των απαιτήσεων τα κράτη-μέλη άλλωστε είναι ελεύθερα να καθορίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα ε, προχωρήσουν προς την κλιματική ουδετερότητα. Η Πολωνία που έχει μεγάλη εξάρτηση χρειάζεται επιτυχημένα εργαλεία προκειμένου να πετύχει τη δίκαιη μετάβαση. Και πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες ε, μορφές ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να έχουμε και φρέσκο χρήμα και όχι μόνο μεταφορά πιστώσεων από την κυνηγιορική πολιτική, για παράδειγμα, ή την πολιτική συνοχής, που είναι τόσο σημαντικές πολιτικές δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση και για την κατανομή και τους διάφορους περιορισμούς. Η Πολωνία πλήττεται βαρύτατα ουσιαστικά θα πρέπει να μεταφέρει χρήματα από τον Εθνικό Προπολογισμό Συνοχής στο Ταμείο Δικής Μετάβασης. Και αυτό θα μπορούσε να αιτιολογηθεί μόνο εάν υπάρξει πάρα πολύ πρόωρο σχεδιασμό των σχετικών δαπανών, δαπανών για το κλίμα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπο με τον οποίο θα διαρθρωθεί αυτό το Ταμείο Δική Μετάβαση και η Δική Μετάβαση. Πρόεδρο, για η τελευταία παρατήρηση. Ο Νίκλας, που έχει ήδη μιλήσει βέβαια μία φορά και έπειτα θα έχει πέντε λεπτά στη διάθεση το κάθε πυρογνώμων σε περίπτωση που θέλει τον λόγο. Α, δεν θέλετε. Πολύ καλά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα αφήσουμε στην Κομισιόν έτσι, πιο πολύ χρόνο για να απαντήσει και εν συνεχεία θα ακούσουμε τις καταληκτικές παρατηρήσεις από τον εισηγητή μας και θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Παρακαλώ. Ναι, θα τα πω γερμανικά τώρα ε, γιατί έχω ένα σχόλιο ε, και κάποια άλλα ε, γενικά σχόλια. Το πρώτο σχόλιο για τον Πρόεδρο, τη Γραμματεία, την Επιτροπή μας. Νομίζω σήμερα ε, είδαμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ έτσι, θερμή ανταλλαγή απόψεων. Αλλά σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η ανταλλαγή, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο και όχι τόσο μονολόγους. Γιατί ενώ ήταν ανταλλαγή αυτή απόψεων, δεν ήταν κάτι πέραν από μεγάλους μονολόγους. Τώρα, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, ε, θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν θέλουμε να μείνουμε προσκολλημένοι όμως στο παρελθόν και να διατηρήσουμε τα πράγματα ως είχαν. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις ε, για το μέλλον και εμείς θέλουμε ως κοινοβούλιο όσο το δυνατόν συντομότερο να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό το έχουμε αποφασίσει. Σε τέσσερις ε, τουλάχιστον περιπτώσεις λέμε εδώ είναι πολύ, εδώ είναι πάρα πολύ κτλ. Όχι. Πρέπει να δούμε πώς θέλουμε να δημορφώσουμε το μέλλον και όχι να κοιτάμε τι γίνεται μέχρι τώρα. Βέβαια έχουν φύγει αυτοί οι συνάδελφοι για τους οποίους, ε, απευθυνόμουν, αλλά ε, επειδή είναι εδώ ο κύριος Μπιζού, ε, να του πω κάτι συγκεκριμένα. Χαίρομαι γιατί μιλήσατε για τις μελλοντικέ τεχνολογίες, γιατί πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε ουσιαστικά περισσότερες εξαγωγές. Έχουμε φωτοβολταϊκά στη Γερμανία. τι κάνουμε με τις εξαγωγές Το 2009 ε, ουσιαστικά ε, πέσανε πάρα πολύ, έπεσε πάρα πολύ η παραγωγή γιατί σταμάτησαν να δίνονται επιδοτήσεις σε αυτό το κλάδο και μέχρι και από την Κίνα εισάγουμε τώρα. Ε, το ίδιο ισχύει με την αιωλική ενέργεια. Οι Σκανδιναβοί φίλοι μας είναι πάρα πολύ καλοί στον τομέα αυτό. Ε, από τις σκανδιναβικέ χώρες δεν βρίσκεις ε, καλύτερες ε, και εξάγονται και προς τις ΙΠΑ και άλλες χώρες του κόσμου. Πρέπει να στραφούμε σε αυτούς που έχουν εμπειρία και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα και για το Σάφο Πέρες πάλι τη συνάλφο που μίλησε για την Αραγών. Υπάρχει και εκεί ένα πρόγραμμα που, από Ευρωπαίους ερευνητές ε, για την παραγωγή υδρογόνου από την ε, ηλιακή ενέργεια. Μην πάμε να αγοράζουμε από την Κίνα. Μπορούμε να τα ε, παράγουμε εδώ. Ε, ούτε από τη Βόρεια Αμερική να εξαρτώμεθα για πολλά πράγματα. Μπορούμε εμείς εδώ να προωθήσουμε νέες τεχνολογίες, μελλοντικέ τεχνολογίες. Και δεν αρκεί να λέμε εδώ έχει πρόβλημα, εκεί υπάρχει πρόβλημα κτλ. Και για την κυρία Κρούκ, για την πυρηνική ενέργεια, γιατί και αυτή αναφέρθηκε. Ακούστε, πρέπει να υπάρξει μετάβαση το συντομότερο δυνατό. Έκλεισε το μικρόφωνο του ομιλητή. Ε, ε, ε, συγγνώμη. Έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο 15 χρόνια γίνεται αυτό το έργο της ανοίξης του τελευταίου πυρικού σταθμού που έχει ανοιχθεί Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, μέχρι το 2050, αν πάμε έτσι, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Μην εστιαζόμαστε πλέον στην πυρηνική ενέργεια. Ας ε, αλλάξουμε. Πρέπει να στραφούμε, παραλαμβάνω, στο μέλλον, στις μελλοντικέ τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Bon, tu les discours. Λοιπόν. Λυπάσαι που έγιναν μονόλογοι, αλλά δεν είσαι και δεν έκανες και εσύ κάτι άλλο. Μονόλογο έκανες. Ε, και ξέρει κάτι, αν δεν έχουμε οργανώσει καλά μια συζήτηση θα επικρατήσει αναρχία. Επίσης, είμαστε συνομοθέτες. Άρα πρέπει να δεχθούμε ότι αυτοί που θα έχουν την ευθύνη και θα πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αφού ακούσαμε τους εμπειρογνώμους θα πρέπει να, λαμβάνουν, να αναλάβουν τι ευθύνε. Ακούσαμε τις απόψεις, ακούσαμε τις ερωτήσεις, ακούσαμε και τις ομιλίες και τους μονολόγους και πολύ καλά κάναμε γιατί είμαστε στην αρχή της εξέτασης αυτού του ταμείου. Είναι πάρα πολύ πλούσια η συζήτηση και νομίζω ότι ως πρώτη ανταλλαγή απόψεων ήταν άκρο ενδιαφέρουσα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις διαφορές στις απόψεις και στις οπτικές γωνίες. Σίγουρα όμω όλοι ε, συμφωνούμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ σοβαρά ε, τον σχετικό κανονισμό. Θα δώσω το λόγο στην... Ε, επειδή μου είπαν ότι η ΕΟΚΕ εκπροσωπείται εδώ, παρακολούθησε τη συζήτηση, δεν το γνώριζα, δεν γνώριζα ότι ήσασταν εδώ, οπότε η εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ θα έχει το λόγο για δύο λεπτά αλλά και με τον σε ΣΕΟΚΕ δεσμεύτηκα ότι θα επανέλθετε, θα επανέλθετε στην Επιτροπή μας ε, για να κάνετε μια πολύ έτσι πιο ενδελεχή παρουσίαση πάνω σε πολλά σήματα, μεταξύ αυτών και Επιταμείου Δίκαιες Μετάβασης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Είμαι ένα αναπληρωματικό μέλος στη δεύτερη ομάδα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ε, δεν θα μακρηγορήσω, γιατί πολλά υπόθηκαν. Εμείς εγκρίνουμε το σχέδιο του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενθουσιοδό μάλιστα, αλλά και εμείς έχουμε κάποια ερωτηματικά για κάποια μέρη, κάποια τμήματα. Καταρχάς, θα θέλαμε αυτό το ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση, να μην περιοριστεί στη χρηματοδότηση έργων απαλλαγή από τις εκπομπές ε, της Ανθρακούχέ, αλλά να κάνει και άλλα πράγματα. Μας ανησυχεί ε, η πιθανότητα να μειωθούν ε, περαιτέρω, η, να μειωθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤΣΙΝ. Ε, θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει μια συνεχής ε, παρακολούθηση, έλεγχος και ε, επαλήθευση του καταμερισμού των πόρων αυτών, οι πόροι δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που όλοι θα θέλαμε. Θέλω να πω ένα μόνο πράγμα, γιατί όλα τα άλλα υπόθηκαν. Ας λάβουμε υπόψη ότι θα έπρεπε να εναρμονιστούν τουλάχιστον κάποιες δράσεις, γιατί ζούμε σε μια διασυνδεμένη παγκόσμια οικονομία. Παραδείγματο χάρη, το κλείσιμο ενός ορυχείου στην Τσεχία μπορεί να έχει σαν συνέπεια η επιχείρηση που παρήγαγε ε, τα υλικά που χρησιμοποιούσε αυτό το ορυχείο που βρίσκεται ας πούμε στην Ολλανδία ή στην Ισπανία ε, να υποστεί τις συνέπειες ε, για παράδειγμα. Δηλαδή ε, Θέλω να πω ότι οι δράσεις που εφαρμόζονται σε μια περιοχή μπορούν να έχουν συνέπειες και σε άλλες περιοχές. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας και τους εργαζόμενους, γιατί οι τοπικές αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν εδαφικά σχέδια. Γιατί αν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, οι εργαζόμενοι αυτοί ούτε θα επανεκπαιδευτούν, ούτε θα αποκτήσουν νέε δεξιότητε, ούτε θα βρουν άλλη θέση εργασία. Με την έννοια αυτή λοιπόν και κατά τον τρόπο θεωρούμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις για τις οποίες ήδη ε, υπάρχει μια κάποια ευελιξία θεωρούμε ότι η ευελιξία αυτή θα πρέπει να αυξηθεί και κατά πολύ μάλιστα. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η λύση που έχουν τα κράτη ε, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες ε, καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. Τέλος, ξέρουμε ότι η φόρος ανάπτυξη, η δράση για το κλίμα έχουν θετικές επιπτώσεις και πραγματικά δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας, σε δραστηριότητες ε, ε, αποκατάστασης, απορρίπανσης κλπ. Ε, αλλά ε, δεν θεωρούμε ότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ε, περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτά είχα να σας πω. Η πρώτη συζήτηση θα γίνει αύριο μεταξύ μας. Ε, προβλέπεται να περάσει από την Ολομέλεια ε, τον Απρίλιο και θα γίνει και μία επίσκεψη μελέτη στη Δυτική Μακεδονία ε, ακριβώς για να ε, δούμε επιτόπου ποιες θα είναι οι συνέπειες του, της πάυσης της εξορρυκτικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στον ή μάλλον να πω στον εισηγητή ότι πρέπει να παραμείνει σε συνεργασία μαζί σας. Η... Το εγχείρημα που προτείνουμε είναι δύσκολο, είναι όμως απαραίτητο. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή για πέντε λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολύ γενναιόδωρο εκ μέρου σα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Πολλά είναι τα στοιχεία που πρέπει να εμπλουτίσουν τη συζήτηση. Θα σταθώ σε δύο-τρία μόνο. γιατί πιστεύω ότι πολλοί μίλησαν για πιο ευρύτερες ε, ε, απόψεις και για την περιβαλλοντική πολιτική και για την εμπορική πολιτική και την ενεργειακή πολιτική. Ε, όλα αυτά δηλαδή ξεπερνούν το θέμα που μας απασχολεί. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω επ' αυτού. Όποτε θέλετε διευκρινήσεις μπορούμε να το δούμε διμερώς. Θέλω καταρχάς λοιπόν να μιλήσω για το ε, δίκαιο χαρακτήρα αυτού του ταμείου, γιατί ασκήθηκαν κριτικές γι' αυτό ασκήθηκαν επικρίσεις. Έχουμε μια κοινή προοπτική μεταξύ Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής. Είναι στραμμένα προς το μέλλον, είναι για δεσμεύσεις που θα γίνουν στο μέλλον. Δεν μιλούμε για ανταμοιβή, για παρελθούσες δράσεις. Θέλουμε να προχωρήσει μια διαδικασία η οποία για να γίνει πρέπει να υπάρχουν διάφορες δράσεις και το ίδιο ισχύει και με την πολιτική συνοχής υπό την έννοια ότι και η πολιτική συνοχή εστιάζει την προσοχή της στις προκλήσεις και οι πόροι δίδονται ε, με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και οι διάφορες ε, περιοχές. Η ίδια λογική μας διέπει εδώ το 30% των πόρων που προτείνονται στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πηγαίνουν στις χώρες συνοχής με ακαθάριστο εθνικό προϊόν που είναι κάτω από το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, θέλω να πω κάτι ξεκάθαρο σε σχέση με τη δικαιοσύνη και το δίκαιο χαρακτήρα του Ταμείου. Το Ταμείο Συνοχής σέβεται πλήρως τους εθνικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η πρόταση αυτή δεν θίγει το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που είναι εφαρμοστέ αυτή τη στιγμή. Το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ε, είναι σε διαδικασία αναθεώρησης και οι κατευθυντήριες γραμμές γίνονται αντικείμενο αναθεώρησης. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία διευκόλυνσης ανακλάδο της οικονομίας τα οποία εξετάζονται και τα εξήγησε το, η ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, δεν έχουμε πρόθεση να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο οι κρατικές ενισχύσεις και θα ακολουθηθεί η ίδια λογική όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή. Τώρα, από πλευράς Ταμείου Συνοχής και σχέσεις του με το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση – Άκουσα τις ανησυχίες αυτές, τις παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, άκουσα τις δύο απόψεις. Ε, κάποιοι ανησυχούν και πιστεύουν ότι το Ταμείο Δίκαιης μας τάβασης κάνει το ίδιο με το Ταμείο Συνοχής και δεν υπάρχει προστιθεμένη αξία. Και από την άλλη ε, υπάρχει εξή ανησυχία ότι το Ταμείο Δίκης Μετάβασης θα κάνει κάτι τελείως διαφορετικό και θα διάσει, θα στραγγίξει τους πόρους από το Ταμείο Συνοχής. Ε, για να σας μιλήσω ειλικρινά. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να γίνει αντιληπτό ως συμπλήρωμα του Ταμείου Συνοχής. Ε, διάφορα στοιχεία του Ταμείου Συνοχής. Στρατηγικές για την έξυπνη εξατομίκευση στοιχεία για την ενεργειακή μετάβαση. Υπάρχουν πολλά τέτοια εκεί. Ε, αλλαγή στις υποδομές για μεγαλύτερη κοινωνική συμπερίληψη. Όλα αυτά υπάρχουν και στο Ταμείο Συνοχής. Εδώ λοιπόν με αυτό το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση πρέπει να διασφαλίσουμε την αλληλοσυμπληρωματικότητα, να έχουμε σωστό πεδίο εφαρμογής. Σας καλώ λοιπόν να αναλύσετε προσεκτικά, να κοιτάξετε προσεκτικά τι προτείνουμε να μπει ως πεδίο εφαρμογής. Υπάρχουν 30 υποτομείς που προτείνονται προς στήριξη και η αποκατάσταση των εδαφών είναι μία από τις 30. Άρα, πρέπει κανείς να εργάζεται με βάση το εφιστάμενο κείμενο για να υπάρχει νομική διάβγεια και ακρίβεια σε αυτά που λέμε. Δεν περιορίζεται το πεδίο εφαρμογή σε οι δράσει που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι η καλύτερη δυνατή χρήση αυτή, δηλαδή πια να είναι ευέλικτο. διαφορετικό διαφορετικές περιοχές, διαφορετικές περιφέρειες, διαφορετικές χώρες ε, αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και από τη στιγμή που περιορίζει κανείς το πιθανό μείγμα πολιτικής περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής ε, τότε θα έχει ένα εργαλείο με αντίκτυπο περιορισμένο, με όχι βέλτιστο αντίκτυπο. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ξέρω ότι μπορείτε να μακρηγορήσετε γιατί σας τέθηκαν πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά οφείλω να σας διακόψω. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είσαστε πολύ ακριβείς στις απαντήσεις σας. Έχουμε τη δουλειά μας, θα την κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τον εισηγητή. Δύο λόγια μόνο, λίγα λεπτά. Ο πρόεδρος θυσιάζεται, ξέρετε όταν ε, δεν ε, διακόπτει τους άλλους. Και εγώ ήθελα να πω πολλά και θυσιάστηκα και δεν θα μπορώ να τα πω. Μανώλη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την άτια οργανωμένη αυτή συζήτηση η οποία μας έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες, μας έκανε πιο πλούσιους σε γνώσεις και ιδέες και είδαμε και διάφορες τοποθετήσεις συναδέλφων για να δούμε πού συγκλίνομαι, πού υπάρχουν διαφοροποιήσεις και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τους ειδικού οι οποίοι μας παρουσίασαν πολλά στοιχεία. Πάνω σε αυτά θα βασιστούμε. Ως πρώτη διαπίστωση βλέπω ότι υπάρχει μια συναντήληψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάμεσα σε αυτά που εμείς έχουμε κατά νου ως συζητητές και οι shadow rapporteurs αλλά και τα μέλη της Επιτροπής της ε, Ρέτζη και αυτό θα μας βοηθήσει στο να διαμορφώσουμε ένα κείμενο που να έχει αυτή τη συναντήληψη καταγεγραμμένη και με συγκεκριμένη θέση που θα μας βοηθήσει και στον τρίλογο και θα βοηθήσει και στις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για να κάνουμε αυτό το μεγάλο όραμα που είναι το Green Deal, την ε, ουδέτερη κλιματική μετάβαση μέχρι το 2050 που δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό το στόχο να είναι μια ευκαιρία και όχι ένα πρόβλημα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Βεβαίως αυτό πρέπει να το κάνουμε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Και αυτά τα πλαίσια είναι δυστυχώς αυτά που συζητούν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα. Αυτό που συζητούν δηλαδή είναι κατά πόσον ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 1,3% όπω λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1,1. Και αυτό μου φέρνει στο μυαλό, ακούγοντα όλε αυτέ τι σημαντικέ απόψει, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε έχουν πολύ μικρότερου και φιλόδοξου στόχου από εμά, σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχουν 6% του ακαθάριστου εθνικού του προϊόντος και εμεί συζητούμε αν θα έχουμε 1 ή 1,3. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να έχω τις, απόψει των συναδέλφων οι οποίοι θα ασχοληθούν με το θέμα Πού θα βάλουμε εμείς το όριό μας. Τα 7,5 δις όλοι λέμε ότι είναι πολύ λίγο ποσό. Το 1 προς 3 που ζητάει η Κομισιόν μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φτάσουμε στο 30% δηλαδή στα 30 δισεκατομμύρια από τα 100 δισεκατομμύρια που θέλουμε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Θέλω λοιπόν και θα έρθω σε επαφή με όλους τους shadow rapporteurs και όλους τους συναδέλφους που μίλησαν να δούμε πού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει αυτό το ποσό να έχουμε μια βασική αρχή, ένα starting point. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ με την άποψη η οποία ακούστηκε ότι αυτό πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία. Ευκαιρία επιχειρηματική, ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο προς τα που πρέπει να πάμε στο θέμα αυτό το ευαίσθητο του περιβάλλοντος και μια ευκαιρία να μην αφήσουμε κανένα πίσω. Για να μην αφήσουμε κανένα πίσω χρειαζόμαστε χρήματα. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να τα βρούμε όχι παίρνοντας από άλλα ταμεία, αλλά από καθαρό χρήμα το οποίο θα είναι αυτή την πολιτική. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω, θα είμαι σε πολύ κλειστή συνεργασία και με εσάς κύριε Πρόεδρε και με τους Προέδρους των άλλων επιτροπών και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών, οι οποίες κάνουν παράλληλα πολύ συγκεκριμένη εργασία. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μα ξεκαθαρίσει ποιε άλλε επιτροπέ και με ποια μορφή θα εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Θα έχετε την υποστήριξη του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής ε, Ρέγγι. Δεν θα πω τίποτε εγώ ε, πάνω σε αυτή τη συζήτηση ε, Έχουμε και άλλες, ε, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Θέλω να ευχαριστήσω απλά όλες και όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτή την πολύ ποιοτική ε, συζήτηση, σε αυτό το εργαστήριο. Θέλω να ευχαριστήσω και το θεματικό τμήμα Β, ε, τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν μέχρι εδώ και έκαναν πολύ ποιοτικές παρεμβάσεις, πολύ χρήσιμες για εμάς στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε ως συνομοθέτες σήμερα. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΟΚΕ, βεβαίω τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ραντεβού αύριο το πρωί 9 το πρωί. Και ευχαριστώ που μείνατε όλοι παρόντες όπως σας το ζήτησα. Ευχαριστώ.